Good morning and welcome to this committee meeting. Uh, we are, I'm very happy. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην πρωινή μας συνεδρίαση. Χαίρομαι διότι βλέπω ότι πολλοί συναδελφοί είναι εδώ παρόντες και αυτό είναι καταπληκτικό. Θα ήθελα να σας πω ότι τα σημεία 14 και 15 γιατί τα ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ε, γνωμοδότηση για τη συνθήκη του Μαρακές θα συζητηθούν περίπου στις 12, 12 και 10. Θα είναι το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης που θα συζητήσουμε. Και έχω και κάποιες ανακοινώσεις να κάνω σε σχέση με τις αποφάσεις των συντονιστών χθες, οι οποίοι ε, δέχθηκαν δύο αιτήματα κατεπήγοντος για αναφορές 1332 και 347 ε, να μπουν στην ημερήσια διάταξη του Ιανουαρίου αντί για του Δεκεμβρίου και η αναφορά για το Σαντιάγο Τέκο Ποστέλα επίσης και κάποια άλλη να μπει στην ε, ημερήσια διάταξη του Ιανουαρίου. Για την αναφορά για το Τάραντο που συζητήσαμε εκτεταμένα πριν από ένα μήνο οι συντονιστές αποφάσισαν να μπει στην ημερήσια διάταξη πριν τη διερευνητική αποστολή, δηλαδή πριν από το δεύτερο εξάμεινο του 2017 όπου προβλέπεται να διενεργηθεί αυτή η διερευνητική αποστολή για να έχουμε ακριβείς πληροφορίες πριν πάμε στο, στο Τάραντα. Η αναφορά 2334 θα μπει στην ε, ημερήσια διάταξη μόλις λάβουμε απάντηση από την Επιτροπή ΕΚΟΝ, γιατί δεν έχει νόημα να συζητήσουμε κάτι χωρίς να έχουμε ακόμα την απάντηση της ενδιαφερόμενης Επιτροπής. Οι αναφορές ε, 337 και 2662 θα μπουν στην ημερήσια διάταξη πριν, ε, αφού τελεσίδικήσουν, πριν βγει, μετά που θα βγει απόφαση δικαστική, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Η αναφορά 8 8-20 θα μπει στην ημερήσια διάταξη του Φεβρουαρίου, είναι του 2015. Και με αυτά λοιπόν εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη του Ιανουαρίου, ενώ για τις εστάσεις που είναι υπό αφισβήτηση, να σας πω ότι οι περισσότερες συμβαστικές λύσεις που πρότεινα έγιναν δεκτές. Όμως για την αναφορά 0626 συμφωνήσαμε να την κρατήσουμε ανοιχτή και να ζητήσουμε πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και υπάρχει ε, και ένα ασφάλμα που διορθώθηκε για την αναφορά 0657, ενώ λεπτομερής κατάλογος των αποφάσεων για τα σημεία που είναι υπό το Β ε, θα ε, συμπεριληφθούν μετά από την ε, συνεδρίαση. Τώρα για τις προετοιμασίες για το Brexit. Είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε επισταμένως. Οι συντονιστές κλήθηκαν να αποστείλουν τα σχόλιά τους αναφορικά με την ανάλυση του αντικτύπου του Brexit. Το σχέδιο που έχει προετοιμάσει η γραμματεία σας έχει διανεμηθεί, το έχετε όλοι και είναι πολύ σημαντικό να το διαβάσετε προσεκτικά και να επανέλθετε στη γραμματεία με τα σχόλιά σας επ' αυτού πριν από τις 8 Δεκεμβρίου, δηλαδή πριν από την επόμενη Πέμπτη. Με αυτά και με αυτά πήγαμε στο ερευνητικό πρόγραμμα και συμφωνήθηκε από τους συντονιστές ε, ότι θα συμπεριληφθούν όλες οι προτάσεις των πολιτικών ομάδων ως μέρη υφιστάμενων προτάσεων ή ως νέα αιτήματα και το Τμήμα Χάραξης Πολιτικής θα οριστικοποιήσει το έγγραφο και η ενημέρωση για την προετοιμασία για την πρώτη σύσκεψη του δικτύου αναφορών έγινε στους συναδέλφους και για αυτή τη νέα διαδικασία σε επίπεδο στελεχών και διοίκηση θα υπάρξει σύσκεψη λίαν συντόμως και η πρώτη συνεδρίαση σε επίπεδο δικτύου θα γίνει στα τέλη Ιανουαρίου μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και τελικά ο Τσιάνι και η Λυπίτα σε πολύ καλή διάθεση. Αυτά έγιναν με τους συντονιστές. Ας προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Όσοι δεν έχετε βάλει την κάρτα στο μηχάνημα, παρακαλώ να το πράξετε. Ο κύριος Μαριάς, έχετε το λόγο. I will be very brief and I will speak in Greek. Ε, κυρία Πρόεδρε, σε σχέση με το report της κυρίας Βαλίνα, Πρώτα απ' όλα να επισημάνω ότι λάβαμε την τελική voting list χτες στις 7 η ώρα το απόγευμα. Έχει υπάρξει μια συμφωνία εδώ να παίρνουμε έγκαιρα τη voting list για να μπορούμε να προετοιμαζόμαστε. Όταν ήμουν ραπορτέρ στην υπόθεση του European Ombudsman την έστειλα τη voting list 24 ώρες πιο πριν για να υπάρχει δυνατότητα στους συναδέλφους να ελέγξουν τη voting list. Υπάρχουν λοιπόν δύο προβλήματα. Πρώτον, στο Compromise 8 και στο Compromise 14. Έχω υποβάλει δύο τροπολογίες, την 172 και την 73. Δεν έχω συμφωνήσει ο CCR να συμπεριληφθεί η τροπολογία μου 172 στο Compromise 8. Δεύτερον, από την voting list προκύπτει ότι η τροπολογία 172 που αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις, εάν γίνει δεκτή το Compromise 8 καταπίπτει. Όμως, στο Compromise 8 δεν περιλαμβάνεται καν η δική μου τροπολογία. Ή δεν υπάρχει έστω και μια αναφορά της δικής μου τροπολογίας και δεν συνήνεσα κι εγώ να υπάρχει αυτή η τροπολογία εκεί. Και στη voting list δεν αναφέρεται καν ότι το ECR είναι στην Compromise 8. Επομένως αυτό το ίδιο ισχύει για μια άλλη τροπολογία, την 73, που αφορά πάλι τις γερμανικές αποζημιώσεις, στο Compromise 14. Επομένως αυτό που ζητώ, και το ζήτησα χτες με email, από την ώρα που έλαβα τη βότην list γύρω στις 7 η ώρα, έπρεπε να την επεξεργαστώ, γύρω στις 9 το βράδυ έστειλα ένα email, ε, θέλω να γίνει χωριστή ψηφοφορία της ε, τροπολογίας 172 και της τροπολογίας 73. Αν το σώμα δεν επιθυμεί, μπορεί να την καταψηφίσει. Αλλά εάν δεν μπουν οι δύο τροπολογίες σε ψηφοφορία χωριστά, τότε ε, δεν δίνεται η ευκαιρία να κριθεί η δική μας τροπολογία. Πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό και είναι αντίθετο με τους κανονισμούς. Και θέλω παρακαλώ να γίνει χωριστά η, τροπολογία, η ψηφοφορία της τροπολογίας 172 και της τροπολογίας 73. Είναι πολύ απλό.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 θα ήθελα να σας δώσω κάποιες ε, συμπληρωματικές πληροφορίες. Ο κατάλογος ψηφοφοριών κυκλοφόρησε όχι στις 11, δεν ξέρω πότε είδατε εσείς τα mail σας, αλλά με ενημερώνουν ότι χθες το βράδυ στις 7 εστάλει. Καλώς. Υπήρξε συμφωνία για τις συμβαστικές προτάσεις από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Εντάξει, όχι από εσά, αλλά ήσασταν μειοψηφία σε αυτή την περίπτωση. Οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες συμφώνησαν κατά πλειοψηφία. Η ομάδα διαπραγμάτευσης συμφώνησε και ως εκ τούτου θα έλεγα ότι οι τροπολογίες ενσωματώθηκαν εκεί όπου μπορούσαν και όποτε μπορούσαν και όταν δεν υπήρχε συμφωνία δεν ενσωματώθηκαν, δεν συμπεριληφθήκαν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα και οι συμβαστικές τροπολογίες δεν χρειάζεται να αφορούν το σύνολο των τροπολογιών, μπορεί να συνεχίσουν να καταπίπτουν τροπολογίες σύμφωνα με τον κανονισμό. Έτσι λειτουργεί κάθε επιτροπή. Δεν θέλω να μπω σε μεγάλη συζήτηση, θέλω ξανά το λόγο για μισό λεπτό. Η κυρία Βαλίνη ζήτησε το λόγο πριν από σας. Καλώς. Καλημέρα σας. Λυπούμε κύριε Μαριά Είχαμε ε, δύο συνεδριάσεις και σε καμία από αυτές τις δύο συνεδριάσεις δεν ε, εμφανιστήκατε. Ούτε εσείς ούτε κανείς από το γραφείο σας. Επομένως είναι αδύνατο να πετύχουμε σε συμφωνίες όταν εσείς δεν συμμετέχετε στις συνεδριάσεις. Και είχαμε δύο συνεδριάσεις. Και όπως είπα, κανείς δεν ήρθε ούτε, ούτε μέλη από το γραφείο σας και το προσωπικό. Επομένως, όταν ολοκληρώσαμε τις συμβιβαστικέ λύσεις στην τελευταία συνεδρίαση στο Στρασβούργο, στείλαμε το προσωρινό κατάλογο την Παρασκευή και μετά από ορισμένες αλλαγές που έγιναν στη συνέχεια, χθες και πάλι 12 το μεσημέρι την ξαναστήλαμε. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνει κανείς είναι να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις για να καταλήγει σε συμβαστικές λύσεις. Προτείνω εσείς οι δύο, λέει η πρόεδρος, παρακαλώ θέλω το λόγο. Συγγνώμη, εγώ έχω το, εγώ έχω το λόγο, λέει ο πρόεδρος, λέει η πρόεδρος. Ναι, αλλά σας τον ζήτησα, το, το ζήτησα. Η πρόεδρος, μπορείτε να το δείτε διμερός. Όχι, πρέπει να το, δεν μπορούμε να το λύσουμε διμερός, αλλά πριν την ψηφοφορία. Θα σας δώσω το λόγο εντός ολίγου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι έχουμε μια πολύ βεβαρημένη μερίσια διάταξη. Δεν θέλω να σπαταλήσουμε χρόνο σε άσκοπες συζητήσεις, αλλά να κάνουμε ε, φοφορία το συντομότερο δυνατό. Κύριε Μαριά. Η τήρηση της δημοκρατίας δεν είναι χάσιμο χρόνο και κάποτε πρέπει να γίνει αντιληφτό σε αυτό το σώμα. Δεύτερον, με τη διαδικασία που προτείνετε εσείς μπορεί να θεωρήσουν τα γκρουπ ότι μια τροπολογία εντάσσεται στο compromise, παρότι είναι τελείως διαφορετική, και με τη συμφωνία της πλειοψηφίας ποτέ μια τροπολογία να μην τεθεί σε χωριστή ψηφοφορία. Και με αυτόν τον τρόπο αφαιρείται το δικαίωμα να τεθεί μια τροπολογία σε ψηφοφορία. Τρίτον, επί της ουσίας, οι τροπολογίες οι δικές μου δεν περιλαμβάνονται στο compromise. Άρα οφείλεται να τις βάλετε σε χωριστή ψηφοφορία. Τέταρτον, για την κυρία Βαλίνα, η τελική λίστα ήρθε στις 7 η ώρα το βράδυ και δεν ήρθε στις 12 η ώρα που λέει. Λοιπόν, εγώ αυτό που ζητώ είναι να γίνουν χωριστές ψηφοφορίες. Αφορούν τις γερμανικές αποζημιώσεις. Βλέπω ότι υπάρχει πλέον αντίθεση από το σώμα στο ζήτημα αυτό, αλλά οφείλετε να το βάλετε σε ψηφοφορία. Δεν μπορείτε έμεσα να καλύπτετε τις τροπολογίες. Okay. Can I just... Καλώς. Πριν δώσω το λόγο στην Άντζελα, να σας υπενθυμίσω ότι μέρος ε, του δημοκρατικού έργου σε αυτό το Νίκο είναι να συμμετάσχει κανείς στη διαπραγματευτική ομάδα και να παρίσταται στις συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Ιδαλλιώς μπορείτε να παραπονιέστε δεξιά και αριστερά στην εισηγήτρια, στην Επιτροπή, αλλά αν δεν είστε παρόν πώς θα μπορέσει να ενσωματώσει οτιδήποτε από εσά αν δεν είστε εκεί. Ούτε οι βοηθοί σα ούτε οι σύμβουλοι πολιτικοί. Ναι, αλλά πρέπει να ακολουθήσετε τον κανονισμό και να βάλετε την τροπολογία σε χωριστή ψηφοφορία. Εάν η πλειοψηφία δεν θέλει την τροπολογία θα καταπέσει. Αλλά δεν μπορείτε να κρύβεστε πίσω από αυτά τα τεχνάσματα για να βάλετε την τροπολογία μου ενσωματωμένη να λέτε και τελικά να μην το κάνετε στην πραγματικότητα. Πρέπει να τη βάλετε σε χωριστή ψηφοφορία. Η κυρία Βαλίνα έχει το λόγο. Λυπούμε πολύ για τα λόγια που ακούω, για το λόγο για τον οποίο ανέφερα προηγουμένως. Δεν συμμετείχατε στις συνεδριάσεις, δεν απαντήσατε σε κανένα mail. Το προσωρινό κατάλογο το στείλαμε την Παρασκευή. Θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει τότε και να πείτε θέλουμε να υπάρξει ψηφοφορία κατά τμήματα τότε από την Παρασκευή. Ε, ας είχατε απαντήσει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα κύριε Μαριά να γίνει ψηφοφορία κατά τμήματα. Εάν το θέλετε το κάνουμε τώρα. Ψηφοφορία κατά τμήματα το 172 και να το πούμε 173. Θα σας παρακαλέσω όμως να συμμετάσχετε εκεί όπου πρέπει να συμμετέχετε. Mr. Marias, there is also a... Κύριε Μαριά, Υπάρχει ένας τρόπος προς τα εμπρός, μου λένε. Μπορείτε να προσθέσετε προφορική τροπολογία και οι συνάδελφοι ή να το απορρίψουν ή να το εγκρίνουν. Είναι μια δυνατότητα. Όχι, είναι διαφορετική ιδέα γιατί έτσι ε, ε, εξαρτάται από τους συναδέλφους να τη δεχθούν την προφορική τροπολογία ή όχι και αυτό είναι τέχνασμα. Εγώ ζήτησα ψηφοφορία κατά τμήματα των τροπολογιών μου. Είναι πολύ εύκολο και παίρνει 10 δευτερόλεπτα. Βάλτε τις δύο μου τροπολογίες σε ψηφοφορία κατά τμήματα σε ξεχωριστή. Θα είχαμε τελειώσει τώρα αν είχατε δεχτεί την πρότασή μου. Πέντε λεπτά συζητούμε τώρα για ένα ζήτημα που θα μας είχε πάρει δέκα δευτερόλεπτα. Καλώς, λέει η Πρόεδρος, ας κάνουμε αυτό σε αυτή την περίπτωση, αλλά ας μην υπάρχει προηγούμενο. Λοιπόν, θα ψηφοφορήσουμε ξεχωριστά την 172 και 207 και θα δείτε τη δημοκρατική διαδικασία. Όχι, είναι 172 και 73. Αυτές είναι οι τροπολογίες. Καλώς, θα τις, ψηφίσουμε ξεχωριστά αυτή τη φορά, αλλά ας μην αποκτήσουμε τη συνήθεια να λειτουργούμε έτσι. Σας καλώ όλους να συμμετάσχετε στη διαπραγματευτική ομάδα και στις συνεδριάσεις. Θα συμμετέχω, αλλά από τη στιγμή που είμαι εισηγητής, όσοι εισηγητή στέλνει κανεί τον κατάλογο ψηφοφορία στο τελικό τι τελευταίε 24 ώρε. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Ακούστε, είναι πολύ νωρί το πρωί. Παρακαλώ, μην χαμαλάτε τη μέρα στου υπολείπου και α προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Okay, let's go. Προχωρούμε. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 107 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Το πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Ας προχωρήσουμε στη συμβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 114 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1-2-2 σε τμήματα επίσης. Το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Άποχες. Θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Αποχές. Θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Βλέπω ότι δεν ψηφίζετε. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ένα 30 τροπολογία υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 1-3-1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1-3-6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1-3-7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1-3-8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1.39 υπέρ κατά αποχές δεν είναι πολύ σαφές, ας το ελέγξουμε. Πέρα στις ε, τροπολογίες απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, θα το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία.

146. Η 146 καταπίπτει. 147 υπέρ. Κατά. εποχές Ελέγχουμε. Εγκρίθηκε. Πάμε σε 148, 149 και 150. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Η 151 έχει αποσυρθεί. Πάμε στα 152 υπέρ. Κατά. Εποχές. Ελέγχουμε την 152. Πέρας ψηφοφορίας συγκρίθηκε 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 156 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 160 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές το ελέγχουμε. Ψηφίστε τώρα. Πέρας φοφορίας. Έχει εγκριθεί. 161 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Την ελέγχουμε. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Σαφέστατα. 163 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείται. 164 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 165 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. Δεύτερο θέμα υπέρ κατά αποχές το ελέγχουμε. Ψηφίζουμε τώρα. Υπέρ ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε χωριστά την 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εμφανώς. Εντάξει, για λόγους δημοκρατίας ελέγχουμε το σημείο αυτό ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. And the vote is closed. Εμφανέστατα έχει απορριφθεί. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 177 Καταπίπτει αυτή. Πάμε στην 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 179 Η 176 έχει απορριφθεί. Η 177 δεν καταπίπτει. Δεν καταπίπτει. Θα πρέπει να ψηφίσετε λοιπόν 177. Ψηφίζουμε την 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 199 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. 191 και 192. Είναι πανομοιότυπες. πέρ κατά, εποχές, απορρίπτονται. 193. Υπέρ, κατά, εποχές, την ελέγχουμε. Ψηφίσουμε τώρα για την 193. Πέρες ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. 194 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για να την ελέγξουμε. Δεν σηκώνετε το χέρι σας όλοι. Εσύ, Μάργαρετ, ναι, αλλά όχι οι υπόλοιποι. Πέρας και έχει εγκριθεί, όντως. Συμβασμός 11 υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 98 υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 201 κατά εποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 και 205 ελέγχουμε χρονικά τη 203 ψηφίσουμε τώρα Απορρίφθηκε. 200. Πού ήμουνα? Στη 204 και στη 205 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 206. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε σε αναφορές. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν σηκώνει το χέρι σας. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Σαφέστατα ε, περνάει. Σας παρακαλώ σηκώνει τα χέρια σας. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές την ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 σε δύο τμήμα, το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά την ελέγχουμε. Πέρας Έχει εγκριθεί. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι ενούσα απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά άποχες την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Περισσοφορίας έχει εγκριθεί 21 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Δεν χρειάζεται να ελέγξουμε αυτή τη φορά συμβασμός 12 υπέρ κατά αποχές την ελέγχουμε αυτήν ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας. Έχει οθετηθεί Τροπολογία 29 και 30 που είναι ίδιες υπέρ. Κατά. Τις ελέγχουμε. Πέρας φοφορίας Απόρρευτηκε. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 πέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 πέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 πέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά ελέγχουμε ηλεκτρονικά 45 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 46 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 208 υπέρ. Κατά. Την ελέγχουμε χρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 και 50 πανομοιότυπες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 52 υπέρ το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Καταπίπτει. Πάμε στις 57 υπέρ. Κατά. Εποχές. Την ελέγχουμε. Πέρες φοφορίες. Γκρίθηκε. 58 υπέρ. Κατά. Εποχές. Γκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε Απορρίπτεται. Κοιτάξτε όμως με τι διαφορά. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. 66 υπέρ. Προηγούμενη καταπίπτει. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Καν... Απορρίπτεται. Συμβασμός 14 υπέρ. Κατά. Α εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε για μία φορά, ούτως ώστε να είμαστε ειρηνικοί μεταξύ μας. Ας ψηφίσουμε την 73 ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας. Απορρίφθηκε. 76 υπέρ. In block. Okay, can we go? Λοιπόν, ψηφίζουμε μαζικά Α, την 76 με 82. Όχι, δεν μπορούμε. 76 πέρα. Κατά. Εποχές. Το ελέγχουμε. Το σημείο αυτό. Το 76 λέει. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Παραλαμβάνουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά εγκρίνεται 82 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 83 σε δύο τμήματα υπέρ το πρώτο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται το άλλο τμήμα καταπίπτει και πάμε τώρα στην 84 πάλι σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά, ποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 υπέρ, σε δύο τμήματα, το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, ποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, υπέρ του δεύτερου τμήματος, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 Υπέρ. Κατά. Δεν σηκώνει τα χέρια σας. Υπέρ της 92. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ.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 και τώρα, ας ψηφίσουμε συνολικά το έγγραφο με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρα ψηφοφορίας. Ομόφωνα Υιοθετείτε. Έβγε. Θαυμάσια αποτελέσματα έχουμε εδώ. and I encourage colleagues and people that are leaving the... Συνάδελφοι, όσοι θέλουν να βγουν από την αίθουσα, γρήγορα και ήσυχα παρακαλώ, για να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Oui. Πολύ καλά. Το 16 λοιπόν είναι η αναφορά 19-21 ε, του 2016 και θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τους αναφερόμενους στην ε, συνεδρία της Επιτροπής Αναφορών. Είσαστε ευπρόσδεκτοι και ελπίζω ότι θα το διαστανθείτε αυτό για το ενδιαφέρον σας και το συμφέρον των πολιτών το ότι προσέρχεστε στην Επιτροπή μας με τα μελήματά σας. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων λοιπόν στην πραγματική ζωή και πραγματικό χρόνο και στο διαδίκτυο ε, μεταδίδεται η συνεδρίασή μας και έτσι λοιπόν με τη δυνατότητα συμμετοχής ακόμα και από απόσταση είναι θετική η προοπτική. Λουίς Ροντάν πρώτα και στη συνέχεια ο Αλέν Ροσντιάν και μετά ο Ιβάν Χότσον. Έχετε μερικά λεπτά, το πολύ πέντε ο καθένας. Πρέπει να είμαστε πολύ ευθυροί με το χρονοδιάγραμμα σήμερα. Έχετε τον λόγο και μπορείτε να διαιρέσετε τον χρόνο αναμεταξύ σας. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Εκπροσωπώ την ε, Ομοσπονδία ε, ε, εμπορίου και υπηρεσίων και την ε, Συνομοσπονδία Εργαζόμενων στη Γαλλία. Εκπροσωπούμε αναφορά για την ε, ε, εργασία την επισφαλή σε τρεις χώρες. Η McDonald's ουσιαστικά εξάγει το αυτό του είδους εργασία στην Ευρώπη για να υπάρχει αβεβαιότητα στο χώρο εργασίας και υποβάθμιση των θέσεων και των συνθηκών εργασίας οι μισθωτοί βλέπουν τη δουλειά τους να γίνεται ακόμα πιο επισφαλής και όλα αυτά αμφισβητούν ε, στη θέμελα τους αριθμούς και τα στοιχεία τα αριθμητικά που δημοσιεύει η επιχείρηση. Οι τρεις αναφορές έχουν ανέβει στο διαδίκτυο πριν από 10 μέρες και 31.000 ε, πολίτες και μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν υπογράψει. Είναι πάρα πολλοί οι Ευρωπαίοι πολίτες όπως βλέπετε που ε, προσυπογράφουν το σύνολο των αναφορών μας. Θα ήθελα να στηρίξω την ε, γαλλική αναφορά για την περίπτωσή μου η οποία υποβλήθηκε για την Ομοσπονδία Εμπορίου και Υπηρεσιών εξ ονόματος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων. Είμαι μισθωτός εδώ και 10 χρόνια σε αυτή την εταιρεία και είναι εξαιρετικά σημαντική. Ξέρετε, οι μισθωτοί στη χώρα μας βιώνουν μια επισφάλεια, μια βεβαιότητα εξαιρετικά περίπλοκη. Για να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η McDonald's έχει franchise περίπου στα 85% των ε, ταχυεστιατορίων της ε, με δικαιόχρηση και τελικά απομονώνουν τους μισθωτούς οι ιδιοκτήτες. Στη Μασαλία ήταν ε, κάποιος που είχε 15 McDonald's και οι μισθωτοί κατάφεραν να κινητοποιηθούν και ε, να ε, κερδίσουν ε, στις εργασιακές τους διεκδικήσεις. Και τελικά τι έκανε η εταιρεία, ξαναπούλησε τα McDonald's σε άλλους ακόμα μικρότερους για να υπάρχουν μόνο μικρά καταστήματα και άρα να μην υπάρχει καμία δυνατότητα για τους μισθωτούς να συγκεντρωθούν, να μπουν σε συνδικάτο, να εκπροσωπηθούν συνδικαλιστικά, να προωθήσουν συλλογικά τα συμφέροντά τους, να έχουν συμμετοχή στα κέρδη, να ε, υπάρχει ε, μερίμνα για την κοινωνική και πολιτιστική τους πρόοδο και, δεν μπορούν... Ε, και τελικά ο κάθε ιδιοκτήτης, ιδιοκτήτης του καταστήματος, μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει. Υπάρχει ένα τεράστιο νομικό κενό στη Γαλλία για το θέμα αυτό και ελπίζουμε η αναφορά αυτή να τύχει στήριξη για να προχωρήσουν τα πράγματα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω για να αφήσω το δικαίωμα σε όλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, να ξέρετε ότι σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία οι μισθωτοί δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κυρίως οι Γάλλοι μισθωτοί και εφιστούμε την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Εάν ασχοληθείτε με αυτό το θέμα της επισφάλειας στην εργασία των εργαζομένων στα McDonald's, αυτό θα είναι μια πραγματική απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον ευρωσκεπτικισμό και θα δείξετε ότι η Ευρώπη υπάρχει και για να προστατεύει τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους. Ελπίζουμε να στηρίξετε την αναφορά μας για να μπορέσουν όλοι να έχουν δικαιώματα αυτά που αναφέρονται στην αναφορά μας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον Αλά Μπέτερμαν. Καλημέρα και ευχαριστώ για τη δυνατότητα να παραστούμε και να παρουσιάσουμε την αναφορά μας. Πρωτού δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Εθνικής Σοσιαλιστικής Ένωσης εργαζομένων στο Βέλγιο. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία ιστορικού χαρακτήρα για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα ποιο είναι το πρόβλημα στο Βέλγιο. Έχουμε μια αναφορά για τις θέσεις απασχόλησης Flexi Jobs, μια νέα νομοθεσία που προάγει την ευέλικτη απασχόληση. Ο μεγαλύτερος εργοδότης παγκόσμια είναι, σημαντικός εργοδότης είναι και σημαντικός στο Βέλγιο στη χρήση αυτών των ε, δυνατοτήτων και πρέπει να πάμε στο 2015 σε αναδρομή για να δούμε με τα 39 εστιατόρια με 3.500 εργαζόμενους της εταιρείας McDonald's και το αναφερόμαστε το 2015 επειδή από πλευράς Επιτρόπου Τίσεν για το νέο πρόγραμμα εργασίας ε, με την πρόσθετη δημιουργία 500 θέσεων εργασίας ε, κάθε χρόνο 500 λέει νέες θέσεις απασχόλησης θα δημιουργούνται και τι γίνεται μετά από μερικά χρόνια έχουν 75 ε, ε, εστιατόρια αλλά δεν έχουν τους εργαζόμενους που είχαν υποσχεθεί διότι αν πάτε στις Βρυξέλλες στην Μπούς ε, ή στο κέντρο στα εστιατόρια αυτά θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι με ευέλικτο χαρακτήρα και αντικαθιστούν τους μόνιμους εργαζόμενους. 55% των εργαζομένων είναι φοιτητές πανεπιστημίων ή σχολείων που είναι σε επισφαλή απασχόληση και δεν έχουν καμιά εγγύηση για το χαρακτήρα της απασχόλησής τους. Και τώρα η μορφή flexi job ευέλικτης εργασίας είναι χειρότερη ακόμα. Δεν υπάρχει σύμβαση. Υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο και σε καλούν να εργαστείς οποτεδήποτε για μια μέρα ή καθημερινά. Ποιο είναι το πρόβλημα για μας. Υπάρχουν παράπονα όσον αφορά την κυβέρνηση διότι οι φορολογούμενοι στο Βέλιο πρέπει να πληρώνουν τα πάντα διότι ένας εργαζόμενος flexi job δεν πληρώνει κοινωνική ασφάλιση σε σχέση με τα όσα ε, λαμβάνει ο μισθό και αυτό είναι το πρόβλημα και οι εταιρείε μόνο 25% φόρων, φόρους πληρώνουν συνολικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας και ελπίζουμε ότι από το ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρώπη θα δώσει εντολές να διακριβωθεί το τι συμβαίνει με τις κακές αυτές πρακτικές διότι βλέπουμε ότι για τους εργαζόμενους ε, του McDonald's και απευθυνόμαστε σε εσά ε, να μας υποστηρίξετε ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα κακοσκήμενα. Για τα τεχνικά θέματα ο Πρόεδρος θα μπορέσει να παρέμβει να σας τα εξηγήσει. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε. Είμαι πρόεδρος ε, του Βελγικού Σοσιαλιστικού Συνδικάτου. Σίγουρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μεγάλο ποσοστό αδήλωτου, αδήλωτης εργασίας σε εστιατόρια στο Βέλγιο. Υπάρχει ένα νέο νομοθέτημα flexi jobs στο Βέλγιο γιατί ήθελαν να αντικαταστήσουν την, εγκα την λειτουργία των ταμείων. Η FlexiJob είναι μια νέα ρύθμιση σε σχέση με τις μηδενικές συμβάσεις, με μέγιστη ευελιξία για τις εταιρείε που θα χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο απασχόλησης και ελάχιστες εγγυήσεις για τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμό για συλλογικέ συμβάσεις που έχουν συναυθεί ήδη και λειτουργούν. Είναι ένα νέο σύστημα που θα έχει πολύ μεγάλη και έχει μεγάλη επίπτωση στην κατάσταση των εργαζομένων, αλλά και σε σχέση και με τον ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών. Θα έχουν τη δυνατότητα, όπως η εταιρεία McDonald's, σε διάφορα εστιατόρια που εκμεταλλεύονται αυτέ τι δυνατότητες να διοργανωθούν, ώστε να ανταλλάσσουν εργαζόμενους μεταξύ δύο εστιατορίων, ώστε να παρακάμπτουν τις νομοθετικέ διατάξεις. Στην ερώτηση υπάρχει μια ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα. Η απάντηση είναι σίγουρα όχι. Έχουμε ένα ήδη υφιστάμενο σύστημα με ευελιξία που χρειάζεται ο τομέας και με σεβασμό των ε, συνθήκων απασχόλησης των εργαζομένων. Σε σχέση με τη σύγκριση των αριθμών όσον αφορά τους ε, απασχολούμενους στο σύστημα με την flexi job με απώλεια απασχόλησης ε, ή με το παλαιότερο σύστημα με εκπεριτροπής εργασία. Το σύστημα δεν είναι μια επιτυχία, είναι ένας τρόπος να αποφεύγουν την κοινωνική ασφάλιση και για την, ε, την πρόθεση του ανταγωνισμού. Εδώ σε σχέση με τις εταιρείε, τα στοιχεία τα οποία έχουμε ε, τα, τα επιβεβαιώνουν αυτά. Σε σχέση με την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους ε, με την απουσία διαλόγου ξεκίνησαν διαδικασίες λοιπόν προσφυγής στο, Ευρωπαϊκό, στο Βελγικό Συνταγματικό Δικαστήριο διότι πρόκειται για κοινωνικό αρνητική διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Έχουμε και τον Ιαν Χότσον επίσης παρόντα εδώ. Καλημέρα σας πρόεδρε. Ιαν Χότσον από πλευρά των, του Συνδικάτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι εξίσου δίνη όπως ακούσαμε και σε σχέση με την κατάσταση στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Σε σχέση με νέους ιδιαίτερα που εργάζονται στο McDonald's και περίπου 90% του εργατικού τους δυναμικού είναι σε μηδενικές συμβάσεις ε, με τις οποίες απασχολούνται και σε σχέση με τη συνειδητοποίηση για κάποιους τρόπους για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι μηδενικού επίπεδου συμβάσεις ε, για να ελέγχονται και να υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζομένων με τους φορολογουμένους που πληρώνουν ε, τους φόρους για αυτή την κατάσταση. Οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν αν θα έχουν εργασία μια μέρα ή όχι όταν εμφανίζονται ή αν θα πρέπει να εργαστούν ε, στην επόμενη εβδομάδα. Και εδώ υπάρχει πραγματικά μια δεινή κατάσταση για αυτούς. Δεν ε, υπάρχει κανένα όφελος σε σχέση με την απασχόληση για παράδειγμα για ώρ, κάποιες ώρες ε, μια εγγύου γυναίκας για παράδειγμα που το έθεσε το θέμα και που αισθάνθηκε ότι θα έπρεπε να είχε μια καλύτερη ανετότερη περίοδο ανάπαυσης. Της είπαν όμως ότι δεν ήταν ικανή να εργαστεί και γι' αυτό δεν θα μπορούσε να εξεταστεί η απασχόλησή της. Η κατάσταση λοιπόν για τέτοιους ανθρώπους είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να πάρουν δάνεια. Δεν μπορούν να πάρουν δάνεια, στεγαστικά δάνεια ή να καλύψουν το ενίκαιό τους ή να πληρώσουν την υποθήκη στα σπίτια τους. Με αυτού του είδους του τους όρους απασχόλησης δεν θα έχουν καμιά προστασία απασχόλησης, ε, κανενός τύπου και ούτε καν θα έχουν πληρωμένες διακοπές επίσης. Υπάρχει πολύ αρνητική διακριτική μεταχείριση και πολλή όχληση, μεγάλα προβλήματα που δημιουργούν δημιουργεί αυτή η κατάσταση για τους εργαζόμενους. Ε, σε σχέση με την, το McDonald's αναγκέρθηκε ότι θα υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδος ε, σε σχέση με την ε, εταιρεία McDonald's για να δουν αν μπορούν δοκιμαστικά να απασχολήσουν για κάποιες ώρες εργαζόμενους σε σχέση με την προσφορά που δίνουν στους εργαζόμενους έναντι των μονίμων συμβάσεων. Οι εργαζόμενοι με τους οποίους μιλήσαμε είτε δεν είχαν καν σταθερές ώρες απασχολήσεων απασχόλησης που να τους προσφέρθηκαν ή έγινε με τέτοιο τρόπο η προσφορά που δεν ήταν σε θέση να δεχθούν τις ώρες που τους προσέφερε ο εργοδότης γιατί δεν τέριαζε αυτό το ωράριο με την κανονική τους καθημερινή ζωή και σε σχέση με την ε, δυνατότητα του να μπορούν να είναι παρόντες ε, αυτά τα χρονικά διαστήματα. Και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ε, και η απέτηση σε σχέση με την κάλυψη των βιωτικών τους αναγκών να μπορούν να εργαστούν και αλλού ή και να έχουν πρόσθετη ε, εργασία για πρόσθετα έσοδα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ε, αναμένεται τώρα σε σχέση με την κατάσταση ότι οι μισθοί θα βρεθούν σε δεινή κατάσταση και θα μειώνονται με μια φθήνουσα εξέλιξη και οι συμβάσεις και η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο καθιστά ακόμα πιο δεινή μετά τις τελευταίες εκλογές ε, αυτή την περιθωριοποίηση εργαζομένων και υπάρχουν πιθανότατα πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι ε, ε, ε, έχουν ε, προσωρινή εργασία και έτσι μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον αριθμό. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τώρα έχουμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Θα λάβετε τον λόγο παρακαλώ. Λούλια Ντεμπέης, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά διαβάσαμε αυτές τις τρεις αναφορές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επιβεβαιώνονται οι τάσεις που βλέπουμε να διαγράφονται στην Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης ε, όσον αφορά την προσωρινή απασχόληση και ελαστική απασχόληση που είναι μια αυξανόμενη αύξουσα, σε αύξουσα τάση στην ε, αγορά εργασίας. Και σε σχέση με τους όρους απασχόλησης ε, που αναφέρονται από τους αναφέροντες μπορεί ίσως ε, να κατανοήσετε ότι η προσωπική μου στάση μπορεί να είναι να δείξουμε κατανόηση. Το θέμα όμως είναι τι θα γίνει με την νομική πλευρά και τα κείμενα. Η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική μεταξύ του κάθε αναφέροντος ε, ε, Δεν βλέπουμε να μπορούμε να κάνουμε πολλά για την πρώτη αναφορά για την κατάσταση στην Γαλλία ενώ για τις δύο άλλες αναφορές, την κατάσταση στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις δύο άλλες αναφορές, θα μπορούσαμε να αναλάβουμε δράση ή εν πάση περιπτώσει να διακριβώσουμε περαιτέρω. Τώρα, για την ε, πρώτη αναφορά, εκείνο το οποίο κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε είναι ότι υπάρχει προφανώς ένα εμπόδιο σε σχέση με το ότι εστιατόρια McDonald's λειτουργούν με άδειες, franchise, από μικροεπιχειρηματίες. Αυτό μπορεί να είναι μια πτυχή που μπορεί να ε, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, όμως μπορεί να είναι και εικονική αυτή η κατάσταση και να υπάρχει ίδιος ιδιοκτήτης σε διαφορετικά ε, εστιατόρια. Δυστυχώς δεν υπάρχει από πλευρά κειμένου η βάση για να μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε αυτήν την κατάσταση. Έχουμε μια οδηγία ε, που ε, υποχρεώνει το ότι θα πρέπει να ενημερώνεται και να διαβουλεύεται η επιχείρηση με τους εργαζομένους όταν όμως γενικά υπάρχουν πάνω από 20 απασχολούμενοι στην ίδια εταιρεία όμως δεν υποχρεώνει αυτό τις εταιρείε να δεχθούν ε, ε, συνδικαλιστική εκπροσώπηση, μεσολάβηση ή επιρροή. Για την κατάσταση στη Γαλλία δεν βλέπουμε κάτι το οποίο να έχει παραβιαστεί και να μπορέσουμε να αναλάβουμε δράση. Όσον αφορά την εικονική κατάσταση, κατά την οποία υπάρχει ένας ιδιοκτήτης με αρκετά εστιατόρια, και όταν υπάρχει η υλοποίηση του κατοφλίου σε σχέση με τις διατάξεις που ισχύουν στην Γαλλία θα μπορούσε να διανοιχθεί ε, μια διαδικασία στο γαλλικό επίπεδο για να καταπολεμηθεί η κατάσταση αυτή ενός ιδιοκτήτη με πολλές επιχειρήσεις, πολλά εστιατόρια. Στο ευρωπαϊκό όμως επίπεδο δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα ε, προσφυγής και έτσι ας, επ' αυτού δεν βλέπουμε δυνατότητα να προχωρήσουμε. Στρέφομαι τώρα στην κατάσταση ως έχει στο Βέλγιο Βέλγιο όσον αφορά το καθεστώς flexi jobs που είναι αρκετά περίπλοκο και σύνθετο ως υπόθεση. Εκεί μπορούμε να βρούμε από πλευράς θεμελίου κειμένων κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω εξέταση του θέματος. Υπάρχει μια οδηγία που υποχρεώνει ουσιαστικά τον ε, ε, εργοδότη να δώσει γραπτά την επιβεβαίωση του στον ε, εργαζόμενο όσον αφορά τους όρους και με το flexi job στο Βέλγιο, με αυτό το καθεστώς η σύμβαση πλέον δεν είναι υποχρεωτικό να έχει γραπτή μορφή και αυτό μπορεί να αποτελεί ένα θέμα επί του οποίου θα θεωρούσαμε ότι υπάρχει επίμαχο ζήτημα. Υπάρχει σε σχέση με τη τους μισθούς τους ε, στο Βέλγιο. Πολλά ε, ε, καθορίζονται γραπτός, όμως εδώ ορισμού οι εργασίες, η απασχόληση flexi jobs είναι διαφορετικές. Δεν είναι υποχρεωτική η γραπτή, ο γραπτός καθορισμός, η περιγραφή της εργασίας και του μισθού. Πράγμα το οποίο σε σχέση με το 91-33 μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβαίνει την ε, οδηγία για γραπτές συμβάσεις. Θα έρθουμε σε επαφή με τις ε, βελγικές αρχές για να υπάρξει αποσαφήνιση επ' αυτού πρώτα άτυπα θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και ε, αν δεν υπάρξει κάποια πρόοδος θα υπάρξουν πιο δεσμευτικές διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Και όσον αφορά στη συνέχεια τους όρους απασχόλησης, ε, όσον αφορά τους απασχολούμενους στο καθεστώς Flexi Job, στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε μια οδηγία για την μερική απασχόληση που η βασική της αρχή είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός ή αρνητική μεταχείριση εκείνων που εργάζονται σε μερική απασχόληση έναντι άλλων. Βλέπουμε εδώ τώρα σε σχέση με συγκρίσιμους εργαζόμενους αν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μια σύγκριση για να δούμε αν υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Θα κάνουμε ε, διακριβώσεις για να δούμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο με τους ε, απασχολούμενους με flexi jobs και αν υπάρχει και επίσης διακριτική μεταχείριση πάλι και όσον αφορά το μισθό και πάλι θα έρθουμε σε επαφή με τις βελγικές αρχές για να αποσαφινιστεί αυτό το θέμα και για να μας δοθούν βεβαιώσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα σε σχέση με την τρίτη αναφορά που έχουμε ενώπιόν μας. McDonald's στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα σημαντικό σημείο αναφέρεται εδώ, το καθεστώς δηλαδή των συμβάσεων απασχόλησης μηδενικού επίπεδου, μηδενικών ορών. Μπορούμε να κατανοήσουμε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν δύο είδη, δύο μορφές ε, απασχολούμενων και υπάρχουν και οι ε, αρρωγοί συνεργάτες. Έχουμε ε, εργαζόμενους με αυτό το καθεστώς και έχουμε και τους λιγότερο προστατευόμενους ε, ε, ε, επικουρικά θα έλεγε κανείς εργαζόμενος. Όμως ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει μια, δεν ισχύει μια τέτοια ε, διαφοροποίηση. Είναι κανείς αυτοαπασχολούμενος ή είναι εργαζόμενος απασχολούμενος. Όσοι δεν είναι αυτοαπασχολούμενοι στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να απολάβουν όλων των δικαιωμάτων που προβλέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο με μια πρώτη ματιά οι απασχολούμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και όσον αφορά τους, το McDonald's είναι απασχολούμενοι υπό τον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από πλευρά ευρωπαϊκού δικαίου. Ιδιαίτερα προστασία μητρότητα για τι γυναίκε. Θα εξετάσουμε περαιτέρω, ειδικά σε σχέση με αυτό το καθεστώ ε, απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα αναλάβουμε τα αναγκαία βήματα και διαβήματα μετά από εξέταση των πληροφοριών που θα μα διατεθούν. Αυτό είναι το έργο που επιτελέσαμε μέχρι τώρα. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Uh, ε, πολύ φιλόδοξο. Πολύ σωστά όλα όσα μας είπε η Κομισιόν. Τώρα δίνω το λόγο στους συναδέλφους. Κύριε Γκέρλινγκ, πρώτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους αναφέροντες και την Κομισιόν για τα σχόλια. Νομίζω ότι αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου από κάθε απόψη. Οι τρεις αναφορές αυτές μπορεί να καλύπτουν μόνο τι περιπτώσει που συμβαίνουν σε τρία κράτη-μέλη. Ο συνολικό πληθυσμό είναι 141 εκατομμύρια των τριών αυτών χωρών. Και είδατε πόσο μεγάλη υποστήριξη υπάρχει στη δικτυακή πύλη για τι αναφορέ από πολίτε. Και μάλιστα και από πολίτε άλλων χωρών, πέρα από αυτέ τι τρει χώρε. Και αυτέ οι συμβάσει επισφαλού εργασία ε, εμφανίζονται όλο και περισσότερο, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε όλο και περισσότερα κράτη-μέλη. Και βλέπετε ότι η εικόνα διαφέρει από κράτος σε κράτος παρόλα αυτά. Υπάρχουν μείζων ερωτηματικά που τίθενται, πέρα από τα τεχνικά θέματα που θέτουν ε, οι μεμονωμένες αναφορές. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον που εστιάζουμε στο McDonald's. Είναι σωστό να πούμε ότι αναγνωρίζουμε ε, εμείς οι ευρωβουλευτές ότι το McDonald's δεν είναι ο μόνος εργοδότης που χρησιμοποιεί τέτοιες συμβάσεις εργασίας. Έχει όμως μια ειδική θέση το McDonald's γιατί είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εργοδοτική εταιρεία στον κόσμο. Έχει επίπτωση λοιπόν το τι κάνει σε αυτή την εταιρική κουλτούρα ε, πέρα από το, τα ωριά της δηλαδή. Επηρεάζει και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Επίσης είναι ένα πολύ γνωστό όνομα το McDonald's. Μια πολύ γνωστή μάρκα. Και τομείς όπως το fast food, ξέρουμε ότι από έρευνες που έχουν γίνει, ότι είναι πολύ πιο δίνουν θέσεις απασχόλησης πολύ πιο επισφαλείς από ό,τι άλλες επιχειρήσεις. Δίνουν λοιπόν επισφαλείς συμβάσεις ε, που έχουν επιπτώσεις σε μεγάλα τμήματα των εργαζομένων, πέρα από τους δικούς τους δηλαδή εργαζόμενους. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρές αυτές οι αναφορές. Γι' αυτό κάτσαμε εδώ και ακούσαμε αυτά που μας είπαν οι εργαζόμενοι στο McDonald's. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για αυτές τις αναφορές, ξεκίνησε η δημόσια συζήτηση και εξ αυτού ε, διάφοροι εργαζόμενοι είπαν την ιστορία τους, την προσωπική τους εμπειρία για το πώς επηρεάζει η εργασία τους, τη ζωή τους και τη δυνατότητα ανάπτυξής τους. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Συνθήκη μας δεσμεύει θεωρούμε ότι θα πρέπει να λέει η συνθήκη ότι πρέπει να βελτιωθούν οι... το βιωτικό επίπεδο και οι συνθήκες ζωής. Είναι μια βασική αρχή αυτή. Και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιος... ποιο είναι. Ενώ υπάρχουν όλο και περισσότερα δικαιώματα εργατικού τύπου, Υπάρχουν όμως όλο και περισσότερες περιπτώσεις, υπενήχθηκε σε αυτές, ε, υπενήχθηκε αυτές τις περιπτώσεις η Κομισιόν, περιπτώσεις με παραθυράκια όπου εταιρείε χρησιμοποιούν και αξιοποιούν αυτά τα παραθυράκια για να υποσκάψουν και να διαβρώσουν τα εργατικά δικαιώματα. Προσοχή, προσοχή. Ξέρετε ότι αλλάζει η μορφή η αγορά ε, εργασίας και βρίσκει τους ε, πιο εποφελείς ε, τρόπους απασχόλησης. Εποφελείς βεβαίως για τους ε, εργοδότες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι συντάκτες μας δίνουν πάρα πολλές λεπτομέρειες για τη χρήση αυτών των συμβάσεων. Είτε είναι συμβάσει μηδενικού ωραρίου, χωρίς δηλαδή καμία ώρα εγγυημένη, είτε είναι ευέλικτες μορφές εργασίας, τα flexi jobs στη Γαλλία. Λοιπόν, τι πρέπει να κρατήσουμε. Καταρχάς, όλες οι μελέτες που έχουν γίνει για αυτές τις επισφαλείς εργασίες δείχνουν ότι αυτό επηρεάζει πολύ αρνητικά την υγεία των ανθρώπων. Υπάρχει ένα ευρύτερο κοινωνικό κόστος από τις καλές πρακτικές απασχόλησης, κακές, συγγνώμη, ε, κακές πρακτικές απασχόλησης και το κόστος αυτό το φέρουμε όλοι μας. Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος άγχους, πίεσης στους εργαζόμενους και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ευρύτερο και όλο και μεγαλύτερο κόστος για την κοινωνία εν το συνόλο της. Η ιδέα των συμβάσεων μηδενικού χρόνου εργασίας ή των flexi jobs είναι κακές. Όχι μόνο δεν πληρώνεις για τη δουλειά που κάνεις, αλλά είσαι και σε αυτοαπασχολούμενο σαν ε, επιχειρηματίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, αυτή η διάκριση ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο, δικαιώματα ας πούμε κτλ. Ή ξέρω εγώ στο βελγικό παράδειγμα, η σχέση με, το, με την κοινωνική ασφάλιση. Ε, υπάρχει, δείχνουν όλα αυτά ότι το κόστος πάνω στην κοινωνία και πάνω στον εργαζόμενο είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το κόστος στον ε, εργοδότη. Υπάρχουν λιγότερα δικαιώματα για τον, εργοδότη και ε, για τον εργαζόμενο συγγνώμη, Υπάρχει οδηγία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μερική απασχόληση και άλλες οδηγίες που μιλάνε για την αρχή της ίσης αμοιβή για ίση εργασία και είτε μιλάμε για πραγματικό μισθό, για την αποζημίωση επίπτωση απόλυσης, για την άδεια μητρότητας και κατά πώς πληρώνεται, για τις πληρωμένες διακοπές, όλα αυτά τα πράγματα θίγονται αυτές τις οδηγίες. Και ένα τελευταίο πιο γενικό σημείο πιο βρετανικό ας πούμε. Εμείς αισθανόμαστε αυτά τα στοιχεία. Ε, κάναμε το ευρωπαϊκό δημοψήφισμα τον Ιούνιο και αυτό είχε καταστροφικές επιπτώσεις στις οικονομικές προοπτικές της χώρας. και το δυναμικό της ε, βρετανικής οικονομίας να αναπτυχθεί. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα μιλήσω κυρίως για τη δική μου περιοχή, που την ξέρω καλύτερα, ψήφισαν έτσι γιατί ο κόσμος θεωρούσε ότι τα πράγματα χειροτερεύουν, γιατί ότι θεωρούσαν ότι η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται για αυτούς, ότι δεν υπάρχει κοινωνική Ευρώπη και ότι δεν εξασφαλίζονται τα εργατικά δικαιώματα. Ο κόσμος θεωρούσε ότι δεν είχε τίποτα να χάσει λοιπόν ψηφίζοντας α, τον Brexit. Και όμως δεν είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε πολλά να χάσουμε. Αλλά η αύξηση του, της δημαγωγίας, ε, του αντιευρωπαϊκού πνεύματος που απασχολεί πολύ αυτή την Επιτροπή, γιατί εδώ ακούμε τις ελπίδες ε, και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων από διαφορετικές χώρες και την πίστη τους για το τι μπορούν ε, κατά τη γνώμη τους να πετύχουν από την Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικά. Εάν θέλουμε να παίξουμε κάποιο ρόλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων, είναι σημαντικό να αντιδράσουμε σε αυτό το αίσθημα που έχουν πολλοί Ευρωπαίοι ότι τα πράγματα χειροτερεύουν. Και οι επισφαλείς εργασίες ε, είναι ένα από αυτά τα στοιχεία που κάνουν τους ανθρώπους να οδηγούνται στη δημαγωγία και στο λαϊκισμό. Κομισιόν, θα ήθελα να απαντήσετε στα συγκεκριμένα ερωτήματα των αναφορών. Αλλά και εμεί ω Επιτροπή Αναφορών μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ξέρουμε ότι αυτό είναι μια, ένα ευρύτερο θέμα. Δεν αφορά μόνο αυτέ τι τρει ε, αναφορέ. Έχουμε όλο και περισσότερε επισφαλεί ε, θέσει απασχόληση. Ξέρετε ότι οι τρει αυτέ αναφορέ διέφεραν κατά τη μεταξύ του. Γι' αυτό προτείνω λοιπόν να δουλέψουμε λιγάκι, να ζητήσουμε να γίνουν κάποιες έρευνες για αυτές τις επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και να λάβουμε να εντάξουμε αυτές τις τρεις αναφορές σε μια μεγάλη δέσμη συναφών αναφορών και να κάνουμε μια ακρόαση για τα θέματα αυτά στο μέλλον. Να γράψουμε στο McDonald's. Υπάρχουν ε, και σε άλλες περιπτώσεις, ε, και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε γράψει κατευθείαν σε επιχειρήσεις και έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες και τις ανησυχίες τις δικές μας, αλλά και των πολιτών, να γράψουμε στο McDonald's να ακούσουμε τι έχει να πει. Γιατί καλό είναι να ακούσουμε την απάντηση του McDonald's. Έχει δικαίωμα να απαντήσει. Θα πρέπει επίση να τη στείλουμε στην Επιτροπή Απασχόληση, να ζητήσουμε την γνωμοδότησή τη ή τη γνώμη τη για το πώ μπορούμε να δώσουμε συνέχεια στι αναφορέ αυτέ. Σα ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μας βοηθήσατε τόσο με την υποβολή προτάσεων και καλώ τους συναδέλφους να υποβάλουν προτάσεις, αλλιώς δυσκολεύομαι να συνοψίσω. Η Ελεονόρα Εύη και η κυρία Στανόκα μετά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η περίπτωση της ε, McDonald ε, είναι η νιωστή απόδειξη της απορρίθμισης των φιλελεύθερων πολιτικών που προοδευτικά κατέστρεψε τις κοινοτικές κατακτήσεις, τα δικαιώματα που, για τα οποία πολεμήσαμε για να τα αποκτήσουμε και που ήταν ας πούμε κληρονομιά της ανθρωπότητας. Έχουμε λοιπόν ξέφρενο ανταγωνισμό στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και αντί να βασιζόμαστε στην ε, καινοτομία προϊόντων και διαδικώσεων ε, με κοινωνική δικαιοσύνη, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, και αντί να γίνουν το έμβλημα ας πούμε, των επιχειρήσεων παγκοσμίων, προ, προτιμούν αυτόν τον ξέφρενο ανταγωνισμό, ε, προτιμούν να συμπιέζουν τα κοινωνικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των Ευρωπαίων ε, εργαζομένων. Μιλάμε για μια κοινωνική σφαγή ε, που θύματα είναι οι πιο ανυπεράσπιστοι. Τα δικαιώματά τους τα οποία δεν θα πρέπει ποτέ να θυγούν. Δεν λαμβάνουμε υπόψη το ψυχολογικό σοκ των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν εφιάλτη της επισφάλειας, ε, της φτώχεια που κρύβεται στη γωνία, την ε, έλλειψη της αξιοπρέπειας των ανθρώπων που μένουν ε, χωρίς φωνή και τελικά χωρίς δουλειά. Τους αναγκάζουμε να μένουν σιωπηλοί για να σώσουν τη δουλειά τους παρά τους ε, όλο ένα και αυξανόμενους ε, κινδύνους και συχνά δεν μπορούν εξαιτία αυτών των θέσεων απασχόληση να αντιμετωπίσουν τα πιο γελία έξοδά του για αυτού και για του οικείου του. Και όμω δεν μπορούν να πάρουν κανένα ρίσκο. Ε, καλό θα ήταν να είχαμε μια κάποια σταθερότητα στη ζωή μα όλοι, ούτω ώστε να αντιμετωπίσει τη ζωή με ηρεμία και σταθερότητα. Εκατομμύρια εργα... εργαζομένων στην Ευρώπη σήμερα δεν έχουν κάτι τέτοιο. Και η βήτα του είναι μια συνεχή κούρσα μετεμποδίων. Ε, μία συνεχής αλληλουχία αδικιών, φόβων, καταχρήσεων στο σύστημα αυτό της επισφάλειας, ε, την, βλέπουν τα παιχνίδια των εργοδοτών που παίζουν με όλα αυτά τα παραθυράκια. Και βλέπουμε ότι οι θεσμοί και οι πολιτικοί τους στηρίζουν. Ε, στηρίζουν φοβερές παραβιάσεις των νομοθεσιών ε, και ακριβώς γι' αυτό δημιουργείται αυτή η αίσθηση εξέγερσης, αυτή η διάθεση ε, αγώνα, εξέγερσης, γιατί θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να αλλάξει η ρότα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, να προστατευτούν πραγματικά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων ε, πολιτών, γιατί αλλιώς θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με, τα, με τις προτάσεις της συναδέλφου. Και να, πάει, να πάνε οι αναφορές αυτές στην Επιτροπή απασχόληση και να γράψουμε στο McDonald's. Νομίζουμε ότι είναι σοβαρότατε προτάσεις, μπορώ να τις συμμεριστώ, ειδικά το να γράψουμε στη McDonald's, για να δούμε τι έχει να μας πει. Και επιπλέον να, μάθει και το McDonald's τι είδου αναφορέ λαμβάνουμε για λογαριασμό της. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, επειδή ήταν πολύ δύσκολη η ψηφοφορία σήμερα το πρωί και η συζήτηση από τους συναδέλφους, δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Και αισθάνομαι ότι είναι δύσκολο να περιμένουν οι αναφέροντες. Παρακαλώ να είστε όλοι εξαιρετικά σύντομοι. Η κυρία Ντανόκα. Ναι, αυτό θα κάνω, γιατί ακούσαμε σαφείς δηλώσεις από τους συναδέλφους Ντάρλιν και Εύη Να σας πω ότι καταρχάς είμαι στην Επιτροπή Απασχόλησης και είμαι μέλος και του δικτύου για την απασχόληση και χαίρομαι για αυτές τις προτάσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να προωθηθεί η αναφορά στην Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά να ξέρετε ότι προσπαθούμε να έχουμε νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά το εργατικό δίκαιο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους υπήρξε το Brexit, ότι δεν είναι αρκετή δηλαδή η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή θεώρησε ότι υπάρχουν παραβιάσεις σε δύο περιπτώσεις, σε δύο χώρες, στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Υπάρχει ευρωπαϊκό δίκαιο, ευρωπαϊκή νομοθεσία, ακόμα και αν είναι εξαιρετικά περιορισμένη. θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες για να δώσει συνέχεια στην αναφορά αυτή. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά. Έτσι ολοκληρώνει το κατάλογο των ομιλητών και μόλις με ενημερώνουν ότι οι αναφέροντες ζήτησαν από την ε, Κέρστιν Χαουάλτ να συνοψίσει την άποψή τους εξ ονόματός τους. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά κατά νότα το όριο. Και στη συνέχεια ε, ενημερώθηκα ότι κάποιος θέλει να αξιοποιήσει αυτή τη συνεδρίαση ως δικαστήριο για να καταθέσει αναφορά. Αυτό δεν είναι δυνατόν, δεν το κάνουμε. Μπορείτε μετά να την υποβάλλετε, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, όχι κατά τη διάρκεια. Καλημέρα σας, είμαι, είμαι η Κάστεν Όβαρτ από την Ευρωπαϊκή ε, Συνομοσπονδία Εργαζομένων στον τομέα των τροφίμων και του τουρισμού στην Ευρώπη. Είναι μια αναφορά που στηρίζουμε απολύτως και ευχαριστούμε την Επιτροπή Αναφορών που άνοιξε αυτές τις αναφορές, τις δέχτηκε και τις κρατάει ανοιχτές γιατί δείχνει ότι Πράγματι, οι πολυεθνικές το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν επισφαλείς θέσει εργασία, να υπονομεύουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και να κάνουν dumping εργασιακό και άλλο. Στηρίζουμε τους αναφέροντες. Έχουμε 31.000 υποστηρικτές αυτής της αναφοράς μέσω ενός ειδικού διαδικτυακού εργαλείου που δημιουργήσαμε και τα εκτυπώσαμε για να σας δείξουμε πόσο τεράστιο είναι αυτό το πακέτο των παρεμβαίνοντων και των συμμετέχοντων που στηρίζουν την αναφορά. Συμφωνούμε απολύτως με τις προτάσεις της UDIT και καλούμε την Επιτροπή Αναφορών να εγκρίνει τις αναφορές αυτές και να συστήσει περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών στα κράτη-μέλη. Στηρίζουμε πλήρως την πρόταση η Επιτροπή Απασχόλησης και η Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση να ασχοληθούν με το θέμα αυτό και σας ευχαριστούμε για τις αντιδράσεις σας. και τη γαλλική περίπτωση και το γαλλικό θέμα θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του ελέγχου του αναλαμβάνοντας τη σύμβαση παραχώρησης ε, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της σχετικής οδηγίας και σχετικών κανονιστικών διατάξεων για να έχουμε ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων και για να έχουμε τριπλό αλφα στην αξιολόγηση της κοινωνικής Ευρώπης, αυτά είναι τα ελάχιστα που μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο, σας συνοψίσω. Χαίρομαι διότι η συνεισφορά των νέων συναδέλφων ήταν εξαιρετικά επικοδομητική. Πρότειναν έναν δρόμο προς τα εμπρός. Χαίρομαι διότι η Επιτροπή εξέφρασε τη βούλησή της να συνεχίσει το διάλογο. Με το Βέλγιο πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή. Θα μπορούσε όμως αυτό να επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει το διάλογο με τις τρεις ενδιαφερόμενες χώρες και να επεκτείνει ίσως το πεδίο εφαρμογής και να δει πώς αυτά μπαίνουν σε ισχύ ή κατά πόσο έχουν εφαρμοστεί όχι σε άλλα κράτη-μέλη. Σημειώνω την επιθυμία των συναδέλφων οι δραστηριότητες αυτές να συνδέσουν χρονικά με τη δράση άλλων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως αυτό πρέπει να το εξετάσουν οι συντονιστές για να μπει στην ημερήσια διάταξη. Άρα παραμένουν όλες οι αναφορές ανοιχτές για να διερευνηθεί με ποιον τρόπο θα προχωρήσουμε. Ε, δραστηριότητες όπως ακροάσεις για παράδειγμα ή μαζί και με άλλες επιτροπές. Και ζητούμε από το Τμήμα Χάραξης Πολιτικής να εξετάσει τα γεγονότα, τα στοιχεία, τα αριθμητικά στοιχεία και για άλλα κράτη-μέλη. Όλα αυτά θα τα πράξουμε και θα πρέπει να στείλουμε επιστολές στα McDonald's, στις ενδιαφερόμενες χώρες και να περιμένουμε για την απάντησή τους και μετά θα κάνουμε το επόμενο βήμα. Όμως η αναφορά θα μείνει ανοιχτή. Μπορούμε αυτό να το κάνουμε. Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και σας ε, εύχομαι καλή συνέχεια. Ε, προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημέρης διάταξης. Παρουσίαση της μελέτης για το Λιντέιν, για το γάμα ισομερές του κύκλο εξανίου και ε, το τμήμα χάραξης πολιτικής που ε, ανέθεσε την εντολή για τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Είναι μια παρουσίαση της έκθεσής μας, της έκθεσης για το Λιντέιν, το Λιδάνιο, ένας οργανικός ρηπαντής που εμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που παραμένει. Σημεία αναφορά είναι τα εξή. Στόχος, στόχος της μελέτης ήταν η χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν μολυνθεί με Λιντέιν, ενημέρωση για τις τεχνικές απορρίπανσης εδάφους και υδάτων, ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές και τη δυνατότητα αποκατάστασης. Διακόπτη, η Πρόεδρος. Όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα να το κάνουν ησύχω για να μπορέσουμε να ακούσουμε την εμπειρογνώμονά μας. Έλεγα λοιπόν ότι στόχος είναι να έχουμε ε, ενημέρωση και για το πώς η ενημέρωση δίδεται για το LinkedIn. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση της έκθεσης, την σύνταξη της σε πέντε κεφάλαια που έχουν συμπεριληφθεί. Έχουμε το πρώτο κεφάλαιο γενικές πληροφορίες για το Λιντέιν, δύο η κληρονομιά του Λιντέιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κεφάλαιο τρία ε, επιλογές απορρίπανσης, περιορισμού της ρήπανσης και αντιμετώπισης αυτής, κεφάλαιο τέσσερα βέλτιστες πρακτικές και πέντε επίπεδο πληροφόρησης που δίδεται για το ε, γάμα ισομερές του εξανίου, το Λιντέιν. Εστάλει ερωτηματολόγιο σε πάνω από 100 εμπλεκόμενους φορείς ε, ε, αντιπρόσωποι και στελέχοι της Σύμβασης της Στοκχόλμη συμπεριλήφθηκαν και λάβαμε έξι απαντήσεις από αυτούς. Εκπρόσωποι των αυτόνομων κυβερνήσεων των αυτόνομων κοινοτήτων της Ισπανίας συμπεριλήφθηκαν. Τρεις αυτόνομες κοινότητες απάντησαν. Έχουμε ε, έναν απαντών από το Πανεπιστήμια, έξι απαντήσεις από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις και τρεις από συμβουλευτικά γραφεία και σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σε γενικές γραμμές μιλάμε για ένα ζήζανι οκτώνο εβραίος φάσματος για γεωργικούς και μη γεωργικούς σκοπούς, το οποίο ε, παραγόταν σε 14 ευρωπαϊκές χώρες από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 70 ή και του 90. Παρενθετικά να πω ότι στη Ρουμανία παραγόταν μέχρι και το 2006. Αυτή είναι η ίδια προσέγγιση που είχε ακολουθηθεί και με το DTT και τα άλλα εντομοκτώνα. Πάρα πολλή παραγωγή ήταν στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ισπανία και τελικά στην Ευρώπη είχαν χρησιμοποιηθεί εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι από τη δεκαετία του 50 μέχρι και το 2000. Σε ό,τι αφορά την παρασκευή ε, του Λιντέιν, να σας πω ότι είναι ένα γάμα ισομερές του εξαχλωροκύκλο εξανίου, με πέντε βασικά ισομερή. Το ισομερές είναι μια χημική ουσία που έχει την ίδια σύνθεση με τις άλλες, όμως η θέση των ριζών σε αυτή την περίπτωση, του χλωρανίου στην περίπτωσή μας, είναι διαφορετική. Το γάμα HCH, το γάμα εξάνιο είναι το μόνο ισομερές με ισχυρές ιζανιοκτόνες ιδιότητες και άρα είναι το μόνο που έχει εμπορικό ενδιαφέρον. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι ο κατασκευαστής η διαδικασία παραγωγής είναι πολύ αναπο, αναποτελεσματική. Ένα τόνος λιντέιν, που είναι η εμπορική ουσία, δημιουργεί 6-10 τόνους αποβλήτων των υπολείπων ισομερών του ε, εξανίου ιδιότητες τώρα. Παραμένει. Και ε, για ζεζανιοκτώνα είναι υποτίθεται καλό αυτό, να παραμένει το προϊόν στο περιβάλλον. Είναι βιοσορευτικό, βιοαθρηστικό, υψηλά επίπεδα έχουν βρεθεί σε πάρα πολλούς οργανισμούς, όχι, όχι στους οργανισμούς που στοχεύουν να εξολοθρεύσει μόνο, αλλά και στα θηλαστικά. Έχει ε, ε, οικοτοξικές ιδιότητες, είναι καρκινογόνο Υπάρχει υποψία ότι είναι διαταράκτης των ενδοκρινών και είναι πολύ τοξικό στους υδατόβιους οργανισμούς. Ε, έχει μεταφορά μεγάλης εμβέλειας, έχει βρεθεί δηλαδή σε περιοχές πολύ απομακρυσμένες από την περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε ή από την περιοχή στην οποία παρήχθηκε είχε παραχθεί. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά. Έως εκ τούτου το 2009 το Λιντέιν ε, συμπεριληφθήκε στο παράρτημα 1 της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους οργανικούς ρήπαντες που επιμένουν και ε, παραμένουν δηλαδή για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα ισομερή α και β συμπεριλήφθηκαν επίσης στο κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλες αυτές οι χρήσεις απαγορεύτηκαν ήδη από το 2008 βάσει του σχετικού κανονισμού για τους οργανικούς ρηπαντές που εμένουν. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν υπάρχει κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα μολυσμένα εδάφη, τα εδάφη που έχουν υποστεί αυτή τη ρηπαση ορισμενα Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν εθνική νομοθεσία για το θέμα αυτό. Η ουσία αυτή συμπεριλαμβάνεται το οδηγία πλαίσιο για το νερό ως μέρος του καταλόγου των ουσιών προτεραιότητας. Ποια είναι η κληρονομιά του λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η κληρονομιά της ουσίας αυτής. Έχουμε πάρα πολλά απόβλητα και απορρίμματα, χιλιάδες τόνους έξαχλωροκύκλο εξανίου που έχουν παραχθεί Αυτά τα απορρίμματα είχαν ε, αποθηκευθεί στα, στους χώρους παραγωγής και διατέθηκαν σε χωματερές, χρησιμοποιήθηκαν για μπάζα στις κατασκευαστικές εργασίες ασφαλτόστρωσης και δημιουργίας δρόμων και έγιναν και αντικείμενο ανεξέλεγκτης διάθεσης και ε, παράνομης απόρριψης. Από εκεί και πέρα, από τις καθημερινές λειτουργίες και δράσεις έχουμε ένα spillover, έχουμε επέκταση και έχει υπάρξει μόλυνση των υδάτων, μόλυνση διαφόρων ε, παραγόντων, γιατί το Λιντέιν μεταδίδεται με τον άνεμο, με τα ε, ε, επίγεια ύδατα και τα υπόγεια ύδατα. Και άρα έχει προκαλέσει εκτεταμένη ρήπανση εδαφών, επίγειων υδάτων και του υδροφόρου ορίζοντα. Σε αυτή την εικόνα βλέπετε ε, τοποθεσίες και μέρη παραγωγής που έχουν εντοπιστεί και είναι ε, μολυσμένα. Αυτά είναι με το κίτρινο αστέρι. Ε, επίσης βλέπετε τις χώρες που παράγουν ή που υπάρχει υποψία ότι παράγουν αλλά δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το συγκεκριμένο χώρο ε, παραγωγής που βρίσκεται και αν πράγματι υπάρχει. Αυτές οι περιοχές είναι με κόκκινο ερωτηματικό στην Ισπανία και στην ε, κεντρική Ευρώπη. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε hot spot Έχουμε ορισμένα μέρη δηλαδή καυτά, γιατί εκεί έχουμε χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αποβλήτων εξαχλωροκύκλο εξανίου και ε, μολυσμένο έδαφος. Χρειάζεται ή έχει εφαρμοστεί η τεχνική απορρίπανση των εδαφών, των επίγειων υδάτων και του υδροφόρου ορίζοντα σε όλα τα κράτη-μέλη, όμως δεν έχουν γίνει εργασίες αποκατάστασης σε όλα τα κράτη-μέλη. Εκκρεμούν όλα αυτά. Βλέπετε εδώ τις, τα προβλήματα. Και ποιε είναι οι δυνάμει λύσει, πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα. Οι επιλογές αντιμετώπισης έχουν συμπεριληφθεί σε πέντε διαφορετικά κεφάλαια. Έχουμε μεθόδους περιορισμού ή καύση, αυτές είναι οι πιο συμβατικέ μέθοδοι. Έχουμε φυσικοχημικές μεθόδους αντιμετώπισης, βιολογικές μεθόδους και δυνατότητα ανακύκλωση. Σε ό,τι αφορά τις συμβατικές μεθόδους αντιμετώπισης του θέματος, οι πιο ευρέως διαδεδομένες μέθοδοι είναι τώρα, είναι η εξόριξη, η διάθεση σε ειδικέ συγκεκριμένες χωματερές, χώροι ε, απόθεσης ε, απορριμμάτων, έχουμε ε, τον τρόπο περιορισμού, την άντληση και αντιμετώπιση και την αποτέφρωση. Το πρόβλημα με την εξόριξη και διάθεση όλων αυτών σε συγκεκριμένους χώρους τα φύση ή εναπόθεση απορριμμάτων είναι ότι δεν λύνεται το πρόβλημα, δεν εξαφανίζονται αυτές οι, αυτά τα συστατικά. Σε κάθε περίπτωση είναι ακριβές επιλογές αυτές γιατί θα πρέπει να γίνει και διαχείριση ε, της, ε, του, του, βασικού εδάφους όπου έχει δεχτεί το Λιντέιν και δεν είναι και οριστική λύση γιατί περιορίζεται με το ορυπαντής, η ρηπογόνος ουσία, αλλά δεν καταστρέφεται. Περνάω τώρα στις φυσικοχημικές με, μεθόδους. Υπάρχουν μέθοδοι που αφορούν το, αφαιρούν αφαιρούν από το έδαφος τον ρήπαντη, θερμική απορρόφηση, εξόριξη από το έδαφος με ενεργό άνθρακα. Είναι υψηλή αποτελεσματικότητα της απόσπασης του ρήπαντη, της αφαίρεσης του από, από το έδαφος, όμως δεν ε, είναι 100% και γι' αυτό υπάρχει και αποτέφρωση στη συνέχεια. Άλλες μεθόδου, μέθοδοι που καταστρέφουν το ρήπαντι είναι η κατάλυση βάσης από χλωρίωση, BDC, η in του χημική χημική οξύδωση, ISCO, η φωτοκαταλυτική διαδικασία, η υποβάθμιση με νανοσωματίδια, με ε, χημική αναγωγή σε φάση αέρια. Πάρα πολλές από αυτές τις μεθόδους έχουν δοκιμαστεί μόνο στο εργαστήριο και έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποβάθμιση του Λιντέν σε ε, ε, εγκαταστάσεις παραγωγής που έχουν μολυνθεί ε, και στην Ισπανία, στην αυτόνομη κοινότητα της Αραγωνίας αλλά και στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Μερικές μέθοδοι δηλαδή έχουν δοκιμαστεί μόνο σε εργαστήριο, κάποιες άλλες από αυτές τις εναλλακτικέ μεθόδους έχουν δοκιμαστεί και επί τόπου. Υπάρχει μέθοδος της υποβάθμισης από τους μικροοργανισμούς, δηλαδή βακτήρια, ε, μύκητες και κάποια μικροάλγη ε, να χρησιμοποιούνται Έχουμε βίο αύξηση, ε, ε, προσθήκη των μικροοργανισμών που υπονομεύουν και υποβαθμίζουν την ενεργή αυτή ουσία. Έχουμε βίο διέγερση, ενίσχυση των συνθήκων στους οποίους θα γίνει η βιοδιάσπαση της ουσίας. Σε κάθε περίπτωση μιλούμε για μελέτες σε κλίμακα εργαστηρίου και έχουν ενίοτε χρησιμοποιηθεί τέτοιου είδους μεθόδοι βιολογικές στις κάτω χώρες και, στις, και στη Γερμανία. Έχουμε και τη φύτο αποκατάσταση. Ορισμένα φυτά έχει βρεθεί ότι μπορούν καλύτερα να διασπάσουν το λιντέιν να γίνει φύτο υποβάθμιση, φύτο διάσπαση. Μιλούμε για την διάσπαση των ριζών. Χρησιμοποιούνται τα φυτά και συμβιωτικά μικρόβια εδάφους για να διασπάσουν τους ρηπαντές στην ζώνη όπου αυτοί εντοπίζονται. Έχουν διενεργηθεί και εκπονηθεί κάποιες μελέτες φυτοεκχύλησης, αλλά δεν έχουν γίνει μελέτες κλίμακας επιτόπου. Σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές μεθόδους, μπορώ να σας πω ότι είναι μια προσέγγιση στέρεη από πλευράς περιβάλλοντος, από πλευράς επιστημονικής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί in situ, επιτόπου, όμως υπάρχουν πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που παρεμβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και είναι πρόκληση να τους ελέγξουμε. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες και έρευνες. Μία άλλη επιλογή για την αντιμετώπιση του θέματος είναι η ανακύκλωση. Το πλεονέκτημα εντό εισαγωγικών είναι ότι έχει περιεχόμενο σε χλώριο 70% το Λιντέιν και θα πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ανακύκλωση αυτού. Ορισμένε εταιρείε ήδη είναι δραστήριε σε αυτό το ερευνητικό πεδίο. Υπάρχει όμω ο κίνδυνο εν σχηματισμού περισσότερων επικίνδυνων ουσιών, δηλαδή διοξινών για παράδειγμα, και χρειάζεται αυστηρό έλεγχο των εκπομπών εάν ακολουθηθεί αυτή η μέθοδος αντιμετώπισης του θέματος. Από τη, τα στοιχεία που έχει συλλέξει η έκθεση βλέπουμε ότι υπάρχουν οι βέλτιστες πρακτικές γιατί έχουμε πολλές και διαφορετικές εμπειρίες σε διάφορες χώρες. Διαφάνεια, ε, κατασκευή ε, της, ε, του χώρου υγειονομικής ταφής στη χώρα των Βάσκων, στο Αργαλάριο. Έχουμε το Ισπανικό Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης ε, Δράσεων κατά των οργανικών ρήπαντων που παραμένουν. Έχουμε απολογισμό για τα πεπραγμένα στη Γερμανία ή στις κάτω στο Αμβούργο μεταξύ άλλων ε, και έχουμε, έχουμε λάβει υπόψη την έκθεση των εργαζομένων. Ε, αυτό για την απορρίπανση του σχετικού εργοστασίου στο Αμβούργο. Στο Μπίτερφελτ στη Γερμανία έγινε παρακολούθηση των, του υδροφόρου ορίζοντα των υπογείων υδάτων και έγινε δειγματοληψία, πάνω από 100 δείγματα ελήφθηκαν για να δούμε ποιοι είναι οι ρηπαντές στα υπόγεια ύδατα, ποιοι θα μπορούσαν να είναι και έγινε μοντελοποίηση της κίνησης των ρήπαντων και του τι απογίνονται, τι γίνονται τελικά. Φτιάχτηκε ένα μοντέλο και στη συνέχεια Έχουμε κάποιες εμπειρίες στις κάτω χώρες, το τουέντε για τον εντοπισμό των τοποθεσιών που έχουν υποστεί ρήπανση. Και δημοσιεύτηκε αυτή η ανακοίνωση στην εφημερίδα για να έχουμε ενημέρωση από τους πολίτες, φωτογραφίες συγκεντρώθηκαν, είχαμε ενημέρωση από διάφορες πολλές και διαφορετικές πηγές. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο πληροφόρησης για το Λιντέιν, οι περισσότερες χώρες μπορώ να σας πω ότι δίνουν πληροφορίες για τα επικίνδυνα χημικά και για τους οργανικούς ρηπαντές που, παραμένουν, αλλά όχι πάντα για το Λιντέιν. Δεν, δεν περιλαμβάνονται στοιχεία οι περιφέρειες που έχουν το χώρους που έχουν ρηπαθεί πολύ από το Λιντέιν συνήθως δημοσιεύουν πληροφορίες και σε διαδικτυακή τοποθεσία και δημοσιεύουν την προσέγγιση που έχουν ακολουθήσει για την απορρίπανση του εκάστοτε εργοστασίου. Να σας πω λοιπόν συμπερασματικά ότι έχουμε χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ε, τόνους λινδανίου και αποβλήτων του έξαχλωροκύκλο εξανίου σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία τα ονομάζουμε καυτά σημεία, hot spot στη ε, Τσεχία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία μεταξύ άλλων. Και ε, Υπάρχει απουσία δράσεων αποκατάστασης, κήτη των ποταμών και γι' αυτό έχουμε ευρία ρήπανση των εδαφών, των υδάτων, επίγειων και υπόγειων υδάτων και του υδροφόν ορίζοντα. Και έτσι αυξάνεται το κόστος αποκατάστασης και απορρήπανσης. Υπάρχουν παραδείγματα ποταμιών που έχουν πληγή. ο Δούναβης για παράδειγμα, ο Βίστουλα, ο Ροδανός, ο Βίστουλας, ο Ροδανός μεταξύ άλλων, έχουν εντοπιστεί προβλήματα ε, στις κήτες της αντίστοιχες των ποταμών. Έχουμε ε, χώρους που έχουν ρηπανθεί με το εξαχλωροκύκλο εξάνιο, 88 που έχουν ρηπανθεί και έχουν πολύ έντονη ρήπανση και θα πρέπει οι πρακτικές ε, αυτές οι πρακτικές της καταστροφής των αποβλήτων Λιντέιν και οι πρακτικές αποκατάστασης του εκάστοτε χώρου και της τοποθεσίας να θεωρούνται οι βέλτιστες πρακτικές και να μην υπάρχει εναπόθεση σε χώρο ανεξέλεκτη διάθεση αποβλήτων ή εναπόθεση σε χωματερή ή γεωνομική ταφή. Δεν είναι αυτές οι βέλτιστες πρακτικές. Και τέλος, η εναποθεση σε χωματερη υγειονομικη ταφη δεν ειναι αυτες οι βελτιστες πρακτικες και τελος η αξιολογηση των ε, χώρων που έχουν ρυπανθεί και η η δυνατότητα να μην έχουμε να, καταστραφούν να, ε, τα εργοστάσια αυτά, να υπάρξει γκρέμισμα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνολικό θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Βέγια. Είναι μια από τις περιπτώσεις όπου ευχόμουν να είχα μελετήσει καλύτερα, να είχα σπουδάσει καλύτερα τα θέματα της χημίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι πολύ δύσκολο, δυσχερές θέμα και είμαστε ευγνώμονες από πλευράς του θεσμικού οργάνου ότι έχουμε τώρα αυτή την πολύ χρήσιμη μελέτη. Τώρα θα έπρεπε να δώσω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως είναι πολύ δύσκολο για μένα να προβλέψω το τι θα μπορούσε να προσθεθεί εδώ σε σχέση με τις ε, ευχαριστίες για τη μελέτη που έχουμε και θα είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση αναφορών. Εσείς επιθυμείτε να παρέμβετε ακόμα από την Επιτροπή. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είσαστε πολύ σύντομοι παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτής της πράγματι πάρα πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης. Θα είμαι σύντομος και θα ήθελα να προσθέσω κάποιες νέες πληροφορίες σε σχέση με αυτά τα οποία ήδη παρουσιάστηκαν περιεκτικά για το Λιντέιν ως πρόβλημα για, που αφορά την μόλυνση εδαφών και περιοχών. Και όσον αφορά τη μελέτη και το, την πληροφόρηση, οι κυριότερες χρήσεις ε, του Λιντέν γύρω στο 2000 ε, ε, όσον αφορά τα φυτοκτόνα και τα παρασιτοκτόνα που παρήγονται και σιγά σιγά έπαψαν να παράγονται και σε σχέση με την ε, κτηνοτροφία και τον τομέα της ε, ε, δημόσιας υγείας. Το 2007 έπαψαν να παράγονται και τώρα ο κατάλογος όσον αφορά αυτές τις ουσίες έγινε το 2009 και στη συνέχεια σε σχέση με τον κανονισμό POPS το 2010 ε, όπου όλες οι παραγωγές ε, προϊόντων που ε, στόχευαν στη διάθεση στην αγορά απαγορεύονται για, με αυτή την ουσία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα αποθήκευση και την αποκατάσταση μολυσμένων εδαφών και περιοχών, ο κανονισμός που απαιτεί από τα κράτη-μέλη να αναφέρουν για σε σχέση με τον κανονισμό POPS που βρίσκονται και τι κάνουν σε σχέση με τα παροχημένα αυτά χημικά που βρίσκονται και τι κάνουν. Με πληροφορίες που έχουμε από τα κράτη-μέλη, δύο κράτη-μέλη ταυτοποίησαν τέτοιου είδους α, ε, ε, στοιχεία σε α, ε, μικρές ποσότητες αποθηκευμένων ουσιών και ξεκίνησε, ξεκίνησαν την καταστροφή και αποκάθαση αυτών. Σε σχέση με τις απαιτήσει ε, του κανονισμού POPS και της ε, αντίστοιχη σύμβασης ζητείται από τα εμπλεκόμενα μέρη να ταυτοποιούν και να εντοπίζουν αυτές τις περιοχές και να ξεκινούν ε, με την αποκάθαση και αποκατάσταση αυτών των σημείων. Τα κράτη-μέλη ανταποκρίνονται σε σχέση με αυτό το αίτημα και βρίσκεται υπό εξέλιξη αυτή η δράση. Το Εθνικό Πρόγραμμα η Δράσης υπό το, τη Σύμβαση της Στοκχόλμης από πλευράς της πρόθεσης του από τα κράτη-μέλη. Τρία κράτη-μέλη γνωρίζουμε ότι ε, αντιμετωπίζουν το θέμα των μολυσμένων χωματερών και περιοχών που έχουν μολυνθεί με Λίντεν και σε σχέση με τα εθνικά προγράμματα δράσης και αποκατάστασης ενημερώνουν για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποκατάσταση ε, περιβαλλοντικά αυτών των ε, σημείων. Εμείς βεβαιώνουμε ότι από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα παρακολουθούνται και θα την χάνουν συνέχεια σε αυτά και σε σχέση και με την αρμόδια Επιτροπή και την συνάντηση που διεξάγεται δύο φορές ετήσια για την ε, παρακολούθηση του τι συμβαίνει και την αποκατάσταση. Η επόμενη συνάντηση της Αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί το Δεκέμβριο θα εγγραφεί και το θέμα αυτής της μελέτης στη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής ώστε να υπάρξει και η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών κατά τη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί το Δεκέμβριο για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Από πλευράς της Επιτροπής έχουμε συνειδητοποιήσει φυσικά ότι υφίσταται μείζον πρόβλημα με τις μολυσμένες αυτές περιοχές και σημεία ιδιαίτερα όσον αφορά τον κανασμό Πόψα και πρόσφατα σε σχέση με την χρηματοδότηση και προαγωγή προγραμμάτων στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζονται από πλευρά μας για να διασφαλιστεί ότι θα, υπάρχει, θα υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι και κονδύλια για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το θέμα της μόλυνσης τέτοιων σημείων ώστε να διασφαλιστεί η αποκατάσταση και αποκάθαση στις περισσότερες ε, ε, χώρες από αυτές το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν το δυναμικό οι χώρες αυτές από πλευρά τους για να διασφαλίσουν ε, να εγγυηθούν την ε, καταστροφή αυτών των ουσιών μέσα από τον κανονισμό POPS. Ευχαριστούμε, λέγει η Πρόεδρος, και μια και δεν έχουμε θέμα αναφορά σήμερα, έχουμε την παρουσίαση μιας μελέτης και όχι αναφορά, τις αναφορές ε, που θα αποτελούν τη βάση για την έκθεση αυτή θα τις κρατήσουμε ανοιχτές και θα τις εξετάσουμε εν ευθέτω χρόνο προτείνω να, αποσταλούν, να, αποσταλεί αυτή η μελέτη στις αρχές που γνωρίζουμε ότι υφίσταται για αυτές πρόβλημα και θα εγγραφεί και το θέμα αναφορών για αυτό το συναφές θέμα προς συζήτηση μελλοντικά. Προχωράμε στο επόμενο ε, θέμα, είναι η 2169 του 14 αναφορά και παρίστανται εδώ οι αναφέροντες και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω σε πέντε λεπτά Μάρτα Μαστόν Κάνοβα και το Λινάρες να μπορέσετε να μας παρουσιάσετε το θέμα αυτό σε πέντε λεπτά. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα εν πρώτα όλα εξ ονόματος ε, της ε, περιοχής της Βαλέθια ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα επικεντρώσω την παρέμβασή μου για την παράβαση της οδηγίας όσον αφορά την ε, στρατηγική για το περιβάλλον, διότι θεωρούμε ότι αυτό έχει προτεραιότητα ως θέμα και σε σχέση με το δίκτυο Natura 2000 έχει ήδη αποστείλει μια τέτοια προειδοποιητική επιστολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Βασίλειο της Ισπανίας ε, σε σχέση με την ε, τροποποίηση ότι ε, σε, χωρίς, κανένα, χωρίς καμιά δημόσια συμμετοχή υπήρξε εδώ η αναθεώρηση των 16 προγραμμάτων. Έτσι περιορίστηκε ουσιαστικά η προστασία που απολά λάμβαναν 320.000 στρέμματα, το 12,39% της επικράτειας της αυτόνομης περιοχής της Βαλένσια. Υπήρξε λοιπόν σε σχέση με το 10-15 της 29 Δεκεμβρίου, χωρίς ε, να υπάρχει προηγούμενη αναγνώριση παραβίασης ευρωπαϊκού δικτύου Τίποτα δεν παρακολεί στο μέλλον ο νομοθέτης ε, από πλευράς ε, ε, Βαλένσια να επαναλάβει τέτοιου είδους πράξεις και σε σχέση και με την παραβίαση της σύμβασης του όρχους. Δεν είναι δυνατόν να παραμένει αδρανής η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί μιας τέτοιας σοβαρής παραβίασης για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον παρουσιάζεται εδώ το φαινόμενο ότι μπορούν να τροποποιούνται οι οδηγίες διαρκώς και μάλιστα με αυθαίρετο ασίδωτο τρόπο. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τροποποίηση αυτών των 16 προ, σχεδίων ε, ε, ταξινόμησης αφορούν το 2014 και 2015 και σε, αυτή την, σε αυτό το διάστημα ήταν δυνατόν να γίνουν αυτές οι δράσεις. Γι' αυτό παρακαλούμε να διατηρήσετε την αναφορά μας ανοιχτή και να υπάρξει δική σας παρέμβαση στο Βασίλειο της Ισπανίας ώστε σε σχέση με προγράμματα που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον να γίνονται πάντα σε σχέση με το σεβασμό της σύμβασης του άρχους και της οδηγίας και σε, για τη δράση που α, καταδεικνύουν την παραβίαση της οδηγίας αυτής είναι μια στρατηγική δράση στρατηγικού χαρακτήρου χαρακτήρα που προάγεται από πλευράς αυτών των πρωτοβουλειών τον Ιούλιο 2014 από την κυβέρνηση της ε, Βαλένθια και ε, έγινε αυτό και ε, υπήρξε προσβολή από πλευράς της απόφασης αυτής και από την Ένωση των Περίκων η διαδικασία του επίμαχου θέματος ε, και που ζητείται η επαρκής εφαρμογή της οδηγίας ε, για το νερό και της οδηγίας ε, για το, για το habitat, για τους βιοτόπους και για την προστασία όσον αφορά το πόσιμο νερό και τους τομείς, δασικούς τομείς που πρέπει να βρίσκονται σε ιδιαίτερη, υπό ιδιαίτερη προστασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ε, πτηνά. Λοιπόν, τούτον λεχθέντον το ε, πρόγραμμα σε σχέση με τους φυσικούς πόρους ε, που ίσχυε μέχρι το Δεκέμβριο 2013 ανέφερε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξουν βιομηχανικές δραστηριότητες σε τέτοιου είδους περιοχές ούτε επίσης επέκταση ε, ε, σχεδίων ε, για την κατασκευή κτηρίων και κατοικιών. Και έτσι σε σχέση με την τεχνική πληροφόρηση που υπήρχε διαθέσιμη η τροποποίηση μέσω του νομοθετήματος χωρίς μελέτη επιπτώσεων και συμμετοχή των εμπλεκόμενων είναι αυτό το οποίο ε, προκάλεσε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι σε σχέση με την Επιτροπή ε, ε, Συμμόρφωσης, σε σχέση με τη Σύμβαση Όρχους, δεν δινόταν ο χώρος που έπρεπε στις οργανώσεις των ενδιαφερομένων και σε σχέση και με την ε, δημόσια αυτή ε, υποστήριξη και από πλευρά ε, του δικαστηρίου της Βαλέσια σε σχέση με τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξε κάποια τροποποίηση εξακολουθεί να υπάρχει αρνητική κατάσταση πράγμα το οποίο δημιουργεί μια πρόσθετη δυσκολία για μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ θα λάβει τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας, Πρόεδρε. Ακούσαμε τους αναφερόμενους και θεωρούμε ότι το αντικείμενο αυτής της αναφοράς είναι διτό όμως περιστρέφεται ουσιαστικά σε σχέση γύρω από την παραβίαση προγραμμάτων και σχεδίων και μια και ακούσαμε από πλευράς των πληροφοριών που δόθηκαν για την ε, οδηγία για τους βιοτόπους για πιθανή παραβίαση των διατάξεων όσον αφορά την διατήρηση αυτών των βιοτόπων και ε, την προστασία ε, ειδών και σε σχέση με την, ε, τις ε, νομοθετικές διατάξεις όσο αφορά το 2013 και τον, ε, το νομοθέτημα για τους προστατευόμενους χώρους και την τροποποίηση όσον αφορά προγράμματα και σχέδια για την προστασία των φυσικών πόρων που όπως κρίνουν οι αναφερόμενοι θα εντασσόταν αυτή η τροποποίηση, τροποποίηση των μέτρων διατήρησης που πρέπει να υφίστανται σε, αυτούς, σε αυτές τις περιοχές και δευτερογενός και όπως έγινε γνωστό από τους αναφερόμενους έχει ε, ε, γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή όχι μόνο για την περιοχή της Βαλένθια αλλά και για το σύνολο της ε, Ισπανικής επικράτειας και ξεκίνησε μια προσφυγή επί παραβάση όσον αφορά το άρθρο 4 και το άρθρο 6 της οδηγίας για τους βιοτόπους habitats και σε σχέση και με την ε, περιοχή, ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου στην οποία εντάσσεται η Βαλένσια έχει σημαντική καθυστέρηση η Ισπανία όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των ε, όρων και διατάξεων για την προστασία των βιοτόπων πράγμα το οποίο συνεπάγεται και την υποχρέωση να υιοθετούνται μέτρα προστασίας που θα είναι ενδεδειγμένα για την προστασία των βιοτόπων και των ε, ειδών ε, χλωρίδας και πανίδας. Σαν συνέπεια τούτου ε, υπήρξαν τροποποιήσεις με βάση αυτό το περιφερειακό νομοθέτημα το 2013 και εντάσσονται στην διαδικασία επιπαραβάση που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για αυτούς ε, τους ε, βιοτόπους ε, και για άλλους συναφείς δεν ανταποκρίνονται τα μέτρα στις απαιτήσει εκείνων που έπρεπε να είχαν ληφθεί. Επισημαίνεται ότι ο κύριος στόχος της αναφοράς είναι η παραβίαση της οδηγίας προγραμμάτων και σχεδίων διότι δεν έγινε αντικείμενο μιας ε, στρατηγικής ε, ε, μελέτης και αξιολόγησης αυτή η πρωτοβουλία. Σε σχέση με τις πληροφορίες που μας διαβιβάζονται σήμερα από τους αναφερομένους, αυτός ο νόμος καταργήθηκε και έτσι λοιπόν φαίνεται ότι έχει αρθεί ο λόγος ύπαρξης αυτής της δράσης. Όμως από την άλλη πλευρά θέλει να επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ενημερώθηκε για το ότι η νομοθετική τροποποίηση υπήρξε αντικείμενο και ε, εκτός αν υπάρξει κάποια αντίφαση, διαφορετική τοποθέτηση επ' αυτού ε, σε σχέση με την προσφυγή όσον αφορά το διοικητικό δικαστήριο της Βαλένσια που είχε διεξαχθεί για την πιθανή ακριβώς ε, ίδια ταυτόσημη παραβίαση των διατάξεων της οδηγίας για την προστασία των σχεδίων και προγραμμάτων. Είναι πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις ε, προσφυγές σε εθνικά δικαστήρια. Όταν υφίσταται μια τέτοια προσφυγή σε εθνικά δικαστήρια ε, σε σχέση με τα θέματα τα οποία αναφέρει η αναφορά, αποφεύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναμειγνύεται στις εργασίες ε, στο έργο του, των εθνικών δικαστηρίων. Γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανέλαβε πρωτοβουλίες σε σχέση με την προσφυγή επί παραβάσει ε, μια και τα εθνικά δικαστήρια είχαν επιληφθεί της προσφύγης στην Ισπανία. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε εξεταστικές δράσεις ε, εφόσον υπάρχει επίμαχο ε, εξελίξει δικαστικό θέμα υπό εξέλιξη και πιστεύω ότι δεν προσφέρει καμιά πρόσθετη αξία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπή ε, όταν τα ε, δικαστήρια ως θεματοφύλακες ε, των διατάξεων και του νομοθετικού πλαισίου δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και όσον αφορά την οδηγία για τους βιοτόπους Habitats, να επισημάνω άλλη μια φορά για την υποεξέλιξη προσφυγή ώστε για όλους τους βιοτόπους και της ε, περιφέρειας της ε, Βαλένσια που δεν έχουν ακόμα καθοριστεί ως, ε, ως προστατευόμενες περιοχές ή αν έχουν αναγνωριστεί ως προστατευόμενες περιοχές δεν τη χάνουν των αναγκαίων μέτρων προστασίας όπως θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Είμαστε πάρα πολύ καθυστερημένοι. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Αλβιόλ για ένα λεπτό το πολύ. Σας παρακαλώ πολύ σύντομα, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να σωψήσει κανείς το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους συντάκτες, τις αναφέρουσες, ε, τις οργανώσεις αυτές που εκπροσωπούν, τις θέσεις που πήραν. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό για όλους αυτούς τους λόγους που ακούσαμε, μιλάμε για 300.000 εκτάρια που για δύο χρόνια ε, δεν ήταν καθόλου προστατευόμενα. Λόγω μιας τροποποίησης που έκανε η κυβέρνηση Βαλένθια στην νομοθεσία, μιλάμε και για φυσικά πάρκα τα οποία δεν προστατεύτηκαν για δύο χρόνια και μέσα σε δύο χρόνια άλλαξαν τελείω, ε, άλλαξε το υπέδαφο, το έδαφο. Ε, παρουσίασαν σχέδια για την οικοδόμηση κατοικιών και κτηρίων κτλ. στην περιοχή του Αλκόη Νομίζω ότι το θέμα είναι αρκούντο σοβαρό και μιλάμε για παραβίαση της οδηγίας 2001 κάθετο 42, ε, γιατί αυτή η τροποποίηση του νόμου έγινε χωρίς συμμετοχή και χωρίς διαβούλευση. Φυσικά, η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει κάτι να κάνει, κάπως να ενεργήσει. Θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση. Εάν μπορείτε να αντιταχθείτε, καλό θα ήταν. Θα ήθελα καταρχήν να στείλουμε μια επιστολή στις αρχές της Βαλένθια, για να μάθουμε εάν η κατάσταση η οποία συνέβη στο Αλκόη έγινε και κάπου αλλού. Αυτά τα δύο χρόνια που δεν υπήρχε προστασία, αν, υπήρχε, αν αφορούσε και, και άλλες περιοχές πέρα από το Αλκόη, ας πούμε, και αν υπήρξαν αλλαγές στη χρήση της, του εδάφους. Και να ζητήσουμε αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο, αυτό το project, να μην προχωρήσει μέχρι να υπάρξει μία ε, νομική επίλυση του θέματος. Επίσης, κάτι άλλο που μου φαίνεται πολύ σοβαρό, είναι να γίνει μία έρευνα πολύ συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν, έχει ε, δεν υπάρχει προσφυγή στην ε, δικαιοσύνη. Μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά την ενέργεια της εταιρείας της ε, La Española. εκεί έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αλλά η αλλαγή της νομοθεσίας Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει γίνει τίποτα για τη δικαιοσύνη. Φυσικά ένας πολίτης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιτύχει ας πούμε, την ανάκληση ενός νόμου ε, πήγε προσφεύγοντας μόνο στα δικαστήρια. Άλλαξε λοιπόν η νομοθεσία και χάρη σε αυτή την αλλαγή της νομοθεσίας δεν μπορέσαμε για δύο χρόνια να προστατεύσουμε αυτά φυσικά πάρκα. Είναι πρόβλημα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Επιτροπή Αναφορών να πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη έρευνα για αυτό το φαινόμενο. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να στραφούμε στι αρχέ τη ε, Βαλένθια, να του ζητήσουμε πληροφορίε και να του ζητήσουμε να σταματήσει αυτό το project, να μην προχωρήσει αυτό το σχέδιο οικοδόμηση. Και να ζητήσουμε επίση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει μια έρευνα. Ευχαριστώ. Θαυμάσια. Δεν υπάρχει κανένας άλλος ε, στο κατάλογό μου. Ε, δίνω το λόγο για ένα λεπτό σε κάθε μία από τις δύο μιλήτρες που κάνουν την αναφορά. Να σας διευκρινίσω ότι η τροποποίηση των σχεδίων χωρίς σεβασμό της 2001-42 έγινε χωρίς καμία αξιολόγηση. Μιλάμε ότι έγινε μέσω νομοθετικής πράξης και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα ως πολίτες. Μιλάμε για ζώνες ειδική προστασίας ε, τροποποιήθηκαν, ε, τροποποιήθηκε αυτή η χρήση των 300.000 εκταρίων και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν είχαμε καμία πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Είναι ξεκάθαρο τι μπορούμε να κάνουμε αυτή την αφορά. Την κρατάμε φυσικά ανοιχτή. Και μια και υπάρχουν δύο ε, ανοιχτές διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η Επιτροπή, να ξεκινήσει απλώς ένα διάλογο με τις αρχές της Βαλένθια. Αυτό που είπε και η κυρία Αλβιόλα είναι, τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είναι να απευθυνθούμε στις αρχές της Βαλένθια να τους πούμε ότι έχουμε ε, εξετάσει ε, εκ νέου αυτό το θέμα, ότι είχαμε μία ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν και με τους αναφέροντες και ότι είμαστε πολύ ανήσυχοι για τα τεκτενόμενα. Τι, πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, ας πούμε, σε αυτόν τον πλανήτη. Να διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους και τον πλανήτη και να μην τους εκμεταλλεύεται. Να πούμε ότι έχουμε σοβαρότατες ανησυχίες και θα πρέπει να απευθυνθούμε στις αρχές το αργότερο όταν βγει η απόφαση του δικαστηρίου για τις ακρεμείς διαδικασίες. Και συνεχεία θα επαναφέρουμε το θέμα και θα το βάλουμε στη μέση διάταξη. Πολύ ωραία. Προχωράμε στο επόμενο σημείο, στην επόμενη αναφορά. Την 513. Έχουμε τον αναφέροντα εδώ. Είναι ο κύριος Τζοβάνι που εκπροσωπεί την Επιτροπή. Έχουμε μία ε, παρουσίαση που θα μας κάνει με διαφάνειες. Έχετε το λόγο για πέντε λεφτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, Ευρωβουλευτές. Μία πολύ σύντομη παρουσίαση θα σας κάνω, γιατί νομίζω ότι η αναφορά που έχετε μπροστά σας θα πρέπει να την καταλάβετε το συνόλο της τι νόημα έχει. Ποιοι είμαστε. Είμαστε μια ομάδα απλών πολιτών που θέλουν απλώς να διαφυλάξουν το φυσικό τους περιβάλλον και κυρίως την προστατευόμενη φυσική περιοχή που βρίσκεται στον ποταμό, α, στις όχθες του ποταμού Τρέμπια. Μιλάμε για μία ε, κοιλάδα δίπλα από τον ποταμό, μια πεδιάδα καλύτερα, που ο Χέμιγουέι έλεγε ότι είναι από τις πιο όμορφες του κόσμου. Ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή ε, ένα project βιομηχανικής ανάπτυξης εκεί για την παραγωγή ασφάλτου σε αυτή την ε, κοιλάδα. Εάν προσέξετε το μικρό χάρτη που σας δίνουμε ε, στη διαφάνεια, αριστερά από το χάρτη υπάρχει ο ποταμός Τρέμπια όχι πάνω από 100 μέτρα από την περιοχή που, θα, που θέλουν να φτιάξουν αυτό το βιομηχανικό, τη βιομηχανική εγκατάσταση, μιλάμε για ένα κομμάτι δίπλα, δηλαδή 100 μέτρα, ούτε καν 100 μέτρα από αυτό το μέρος υπάρχει ε, μια περιοχή που προστατεύεται από το Natura 2000. Λοιπόν, με το πρόγραμμα αυτό τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν ε, να φτιάξουν ε, πολύ σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και θέλουν να εγκαταστήσουν και ένα εργοστάσιο ε, εργοστάσιο παραγωγής ασφάλτου. Και πρόσφατα, μάλιστα, προσθέσανε να, και το αίτημα τους δοθεί ε, μία άδεια για την ε, επεξεργασία αδρανών αποβλήτων, δηλαδή αποβλήτων που δεν είναι επικίνδυνα. Εκεί. Μιλάμε για ένα βιομηχανικό πρόγραμμα ανάπτυξης. Και αυτό γίνεται χωρίς καμία, ανα... Ε, χωρίς καμία ε, μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Το πρόγραμμα αυτό, τεχνιέντος πώς, διαιρέθηκε σε μικρά-μικρά κομματάκια για να παρακαμφθούν καταρχάς οι σαφέστατες ενδείξεις που έχει δώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την οδηγία του 2011 κάθετος 92 Επιπλέον, να προσθέσουμε ότι η συμμετοχή των πολιτών σε αυτές τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων δεν υπήρξε. Υπήρξε μηδενική συμμετοχή. Όλες οι παρατηρήσεις των πολιτών, όλες οι προτάσεις ε, που απευθύναμε στους αρμόδιους φορείς αγνοήθηκαν εντελώς και δεν ελήφθησαν ουδόλως υπόψη. Εμείς δεν λέμε ένα όχι απόλυτο στην βιομηχανική ανάπτυξη. Δεν θέλουμε να υπάρξει βιομηχανική ανάπτυξη μη βιώσιμου χαρακτήρα. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη όταν... Να μην λάβουμε υπόψη ότι αυτή είναι μια ειδική περιοχή όπου θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια ε, περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Ούτε μία από, τα, από τις διατάξεις που προβλέπονται στις διάφορες άδειες για τη μετρίαση των επιπτώσεων στο περιβαλλοντικό στο περιβάλλον, συγγνώμη, δεν έχουν υλοποιηθεί. Αντίθετα δίνονται νέες άδειες για νέες εγκαταστάσεις. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι κυρίως απαράδεκτο το να κατακαιρματίζει κανείς project, σε μικρότερα project, σε μικρότερα προγράμματα, προγράμματα που στην πραγματικότητα είναι ένα και μόνο και αδιαίρετο. Γίνεται αυτός ο κατακαιρματισμός, αυτή η διαίρεση, ούτω ώστε να παρακαθούν διάφορες επιταγές, ας πούμε. Καταρχάς, αυτό της περιβαλλοντικής επίπτωσης, δηλαδή της μελέτης περιβαλλοντικού αντικτύπου. Τι ζητάμε από την Επιτροπή Αναφορών. Ζητάμε να κρατήσετε ανοιχτή την αναφορά για δύο βασικούς λόγους. Καταρχάς, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν δύο αρχές απαραβίαστες. Η μία είναι αυτή τη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που λαμβάνονται και που επηρεάζουν το δικαίωμά τους στην υγεία και στη διαφύλαξη του περιβάλλοντός τους. Και δεύτερον, η αρχή εξίσου απαραβίαστη ότι μέσω τεχνητών κατακαιρματισμών ενιαίων προγραμμάτων να παρακαφθούν ξεκάθαρες επιταγές ε, και διατάξεις της ε, Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Νομίζω ότι είναι δύο βασικές ε, αρχές, επί των οποίων δεν χωρεί καμία διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή γίνουν αυτές οι αξιολογήσεις. Νομίζω ότι κανένα δεν θα μπορεί να έχει αντίρρηση. ότι το σχέδιο έχει υποστεί σοβαρή ανάλυση, έχουν γίνει σοβαρέ μελέτες αντικτύπου κτλ. Και άρα αναλόγως μπορούμε να προχωρήσουμε. Μιλάμε για το θέμα του προβλήματος τη της ανάκτησης μη επικίνδυνων αποβλήτων που για να γίνει αυτή η προσπάθεια, δηλαδή ανάκτηση και όχι περαιτέρω κατανάλωση, προχωρούμε σε σε επέκταση ουσιαστικά εγκαταστάσεων, σε επέκταση υπογείων χώρων για να μπορέσει να γίνει αυτή η ανάκτηση. Μου λέτε πώς θα, μπορέσουμε να προβούμε στην ανάκτηση όταν αντίθετα επεκτείνεται τη χρήση υπογείων χώρων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσιπριάνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το εργοστάσιο ασφάλτου υποτίθεται ότι ε, είναι εγκατεστημένο εκτός από ένα χώρο Natura 2000 που εντάσσεται στην οδηγία για τους βιοτόπους πτηνών είναι εκτός αλλά κοντά η οδηγία δεν απαγορεύει τέτοιου είδους δραστηριότητα εντός και εκτός του δικτύου Natura στο βαθμό που τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι συμβατές με τη διατήρηση των οικοτόπων, βιοτόπων και ειδών που εντάσσονται σε αυτή την οδηγία ε, όταν δεν διακυβεύεται η ακαιρεότητα δηλαδή αυτών των περιοχών. Με βάση τα έγγραφα που έχουμε λάβει με αυτή την αναφορά δεν φάνηκε στα σαφή στοιχεία παραβίασης και παράβασης κανόνων και διαδικασιών έτσι όπως προβλέπονται από την οδηγία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οδηγία περιβαλλοντικού αντικτύπου, εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα ήθελα να υπενθυμίσω το εξή: Τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα 2 της σχετικής οδηγίας συμπεριλαμβανομένων διαφόρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων είναι έργα για τα οποία οι εθνικές αρχές πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσο χρειάζεται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη σχετική απόφαση οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τα κριτήρια που απαριθμούνται στο παράρτημα 3 της οδηγίας και τα εν λόγω κριτήρια συμπεριλαμβάνουν επίσης ενδυνάμιση, σόρευση, άθρηση, ε, με την ενέργεια και εφαρμογή άλλων έργων, καθώς και ενδυνάμει η χορύπαση και φωτορύπαση. Είδαμε ότι οι περιβαλλοντικές αρχές σε περιφερειακό επίπεδο εξέφρασαν θετική γνωμοδότηση για το έργο αυτό. Οι σχετικές αρχές ε, το εξέτασαν και θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται πλήρης εκτίμηση, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Άρα σε αυτό το στάδιο δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε σαφή παράβαση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ωστόσο θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι οι εθνικές διοικητικές και δικαστικές αρχές των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με την υλοποίηση και εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών είναι αυτές που είναι και υπεύθυνε που έχουν την ευθύνη να επαληθεύσουν σε κάθε περίσταση και σε κάθε περίπτωση ενδυνάμει κατάσταση μη συμμόρφωσης με τις σχετικές οδηγίες. Οι σχετικές αρχές, επαναλαμβάνω, έχουν και τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες εάν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Οι αναφέροντες έχουν ασκήσει διώξεις, έχουν ασκήσει ένδικα μέσα ενώπιον της Ιταλικής δικαιοσύνη και διεκδικούν και ισχυρίζονται μεταξύ άλλων ότι οι διαδικασίες αδειοδότηση δεν σεβάστηκαν τους σχετικούς κανόνες βάσει ε, της οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν έχουμε όμως ενημερωθεί για την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου συμπεραίνουμε ότι παραμένει εκρεμής. Ως εκ τούτου δεν επιθυμούμε να παρέμβουμε με μια ενεξελίξη εθνική ε, δικαστική διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι έχουν το λόγο. Ελεονόρα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα έργο για το οποίο μας έστειλαν πολύ υλικό οι αναφέροντες και μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε, να δούμε πολύ ξεκάθαρα ποια είναι η κατάσταση της βιομηχανικής αυτής της περιοχής για τον οποίο μιλάνε οι αναφέροντες. Πολύ συχνά προσπαθούμε Προσπαθούν κάποιοι να παρακάμψουν τους κανόνες και να φτιάξουν βιομηχανικά έργα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις γιατί δεν και καλά έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να γίνουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ε, χρησιμοποιούν λοιπόν αυτά τα κόλπα, αυτά τα τερτύπια που καταγγέλθηκαν, προκειμένου να εγκριθεί ένα βιομηχανικό πρόγραμμα. Τι κάνουν λοιπόν. Μιλάμε, Διαιρενού, διαιρούν ένα project το οποίο έχει ενιαίο χαρακτήρα σε μικρότερα project και τα εγκρίνουν βαθμιδών. Μέσα σε μια μεγάλη χρονική διάρκεια. Όλα αυτά τα ήξερε ο Δήμος μέχρι το 2011 και ξέρει πολύ καλά ότι τα διάφορα έργα που εγκρίνονται βαθμιδών είναι τμήμα ενός μεγαλύτερου ενιαίου έργου. Πρέπει να πάει κανείς στα περιφερειακά και εθνικά δικαστήρια για να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα των κατακαιρματισμένων μελετών αντικτύπου που έγιναν και δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσα σε αυτά τα χρόνια. Επίσης υπάρχουν αποφάσεις και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καλούν τις Ιταλικές αρχές να αρχίσουν άπλετο φως και να σταματήσουν αυτές τις πρακτικές. γιατί είναι ασύμβατες με την οδηγία ΕΠΕ. Επίσης είναι ασύμβατες με την ανάπτυξη μιας περιοχής. Πώς αποφασίζουμε να κάνουμε κάποια πράγματα σε μια περιοχή χωρίς την παραμικρή συμμετοχή των πολιτών που ζουν εκεί. Είναι ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που εμείς, ε, η Επιτροπή Αναφορών, ε, το έχουμε δει σε πολλές αναφορές. Είναι μία κραυγή, ένα κόδωνας κινδύνου. Θα πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Θα πρέπει φυσικά να γράψουμε στις τοπικές αρχές για να μας μιλήσουν και να λογοδοτήσουν για αυτές τις πρακτικές. Και φυσικά να καλέσουμε και τους πολίτες να προσφύγουν στα κατάλληλα δικαστήρια. Καλό θα ήταν και εμείς να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κατάλληλα εργαλεία, ούτω ώστε να δούμε και να επαληθεύσουμε αν υπάρχουν παραβιάσεις. Αυτό είναι, εμείς θεωρούμε με βάση αυτά που υπόθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά καλό είναι να ακολουθήσει αυτή η δικασία το δρόμο της στα εθνικά δικαστήρια για να αποδειχθεί. Εξαιρετικά. Και τώρα ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ομιλητών. Ε, έρχομαι σε εσά κύριε Τζιοβάνι. Σας δίνω το λόγο για τις τελικές σας παρατηρήσεις. Ε, σας ευχαριστώ. Να επιβεβαιώσω ότι αυτό το πρόγραμμα, αυτό το project, αυτά τα έργα στην πραγματικότητα εντάσσονται σε ένα πλαίσιο, είναι ένα και ενιαίο. Και αυτό το δείχνουν τα έργα, ε, τα στοιχεία που σας παρουσιάσαμε. Ήταν ξεκάθαρο αυτό ήδη από το 2011 από το 2011 ξέραμε πολύ καλά τι θα γινόταν στην περιοχή. Βέβαια το αγνούσαν οι πολίτες, αλλά οι αρχές το ξέρανε. Και μέσα σε πέντε χρόνια, το 2011 μέχρι σήμερα, δόθηκαν τέσσερις διαφορετικές άδειες. ούτω ώστε να εγκρίνουμε τμηματικά τα επιμέρους τμήματα ενός συγκεκριμένου project, ενός συγκεκριμένου έργου. Ευχαριστώ πολύ. Επομένως ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και μας είπε ότι δεν μπορεί να κάνει και πολλά αυτή τη στιγμή γιατί είναι εν εξελίξει η δικαστική διαδικασία ε, επιτόπου ε, στην Ιταλία για το θέμα αυτό. Όμως από πλευράς δικής μας Επιτροπής μετά από αυτή την ακρόαση μπορούμε να αποστείλουμε μία επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιταλίας και στις τοπικές αρχές στην οποία θα σημειώνουμε ότι αυτό το θέμα μας ενδιαφέρει και μας ανησυχεί. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε την αναφορά μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας για το θέμα αυτό. Αυτό προτείνω. Συμφωνείτε? Καλώς. Έτσι κάνουμε, έτσι θα πράξουμε λοιπόν και ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τζιωβάνι για το ταξίδι του στις Βρυξέλλες. Ε, καλή σας επιστροφή στην Ιταλία. Προχωρούμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μιλούμε για την αναφορά 513 που συνυπογράφουν μισό λεπτό, μισό λεπτό λέει η Πρόεδρος, στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης, το οποίο θα εξετάσουμε τώρα, εντάσσονται διάφορες αναφορές. Ο κύριος Γούτε Βαν από τη Life International που εκπροσωπεί τον αναφέροντα. Έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα παρουσιάσω εξ ονόμως της ε, φρύλα της Βουλγαρίας την αναφορά που υπέβαλαν για τις ανεμογεννήτριες στον πάλσι και στη Καλιάκρα στη Βουλγαρία. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να στηρίζονται, αλλά όταν γίνονται με τη σωστή τεχνολογία και στα σωστά μέρη. Έχουμε ανεμογεννήτριες στην Καλιάκρα. Και αυτή είναι μια σαφέστατη περίπτωση όπου να ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια σε λάθο μέρο. Είναι μια χερσόνησο αυτή η Καλλιάκρα, η χερσόνησο τη Καλλιάκρα, στην παράκτια περιοχή της Βουλγαρία, με πάρα πολλέ δραστηριότητε. Έχουμε πάρα πολλέ αναμογεννήτριε εκεί που χτίζονται και κατασκευάζονται. Εκτό από αυτό, έχουμε και άλλα στοιχεία περιβαλλοντική καταστροφή, γήπεδα του γκολφ που έχουν επίσης χτιστεί και έχουν γίνει αλλαγές της χρήση γης, αλλαγές στη στη γεωργική δραστηριότητα και ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στο περιβάλλον και στην τοποθεσία προέρχεται σε κάθε περίπτωση από τις ανεμογεννήτρες οι οποίες έχουν υποβαθμίσει την περιοχή. Έχουμε αναλάβει πάρα πολύ δράση για να αποφύγουμε τους κινδύνους για τα πτηνά από τις ανεμογεννήτρες. Έχουμε υποβάλει ε, παράπονα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχληση δηλαδή, και τελικά η Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2016 κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δώσει εξηγήσει για την υποβάθμιση της περιοχής και ζητούμε τώρα να μάθουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των πληγήσεων περιοχών και του τοπίου. Βλέπετε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια και πράγματι η κατάσταση έχει βελτιωθεί στη Βουλγαρία με την ενέργεια, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, τώρα η προσέγγιση της χώρας αυτής είναι πιο σόφρονα θα έλεγα. Ε, υπάρχουν χαρτές ευαισθητοποίησης, χαρτογράφηση ευαισθησιών όπου αναφέρεται πού μπορεί κανείς να εγκαταστήσει τις ανεμογεννήτριές του και έχουμε καταλάβει και καλύτερα στη Βουλγαρία τον αντίκτυπο, το θετικό αντίκτυπο των πτηνών τα οποία παρεμποδίζονται από τις ανεμογεννήτριες. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν πολλές οι ανεμογεννήτριες εκεί και καταστρέφουν το τοπίο. Έχουμε τρεις ε, μεγάλες συστάδες ανεμογεννητριών που ε, κατασκευάζονται τώρα και που σκοτώνουν τα πουλιά που ακολουθούν ακριβώς αυτή τη μεταναστευτική οδό από την Αφρική στην Ευρώπη ζητούμε τη βοήθεια της Επιτροπής των Αναφορών για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Βλέπετε εδώ κάποια από τα πράγματα που γίνονται, κάποια από τα πράγματα που κάνουν οι ανεμογεννήτριες. Βλέπετε πόσο συχνά ε, ε, χτυπάει η έλικα της ανεμογεννήτριας πτηνά, στα ε, σταυραετούς, γεράκια, ε, πτηνά τα οποία πετούν αργά και δεν κάνουν πολύ ευέλικτες κινήσεις και τελικά υφίστανται το πλήγμα της εκάστοτε λεπίδας της γεννήτριας, της έλικας. Πάρα πολλά πουλιά βλέπετε ότι πετούν γύρω από αυτές, σαφέστατα γίνεται ζημιά. Τι ζητούμε Θέλουμε η κυβέρνηση της Βουλγαρίας να αναλάβει δράση. Θέλουμε να σταματήσει η ανέγερση ανεμογεννητριών γιατί συνεχίζουν να τοποθετούνται και να καθίστανται ανεμογεννήτριες παρά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θέλουμε να ακυρωθούν οι άδειες λειτουργίας των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες και να αφαιρεθούν κάποιες ανεμογεννήτριες που είναι πολύ εύκολο να αφοβλιστούν και να τοποθετηθούν κάπου αλλού. Είναι σε τόσο λάθος σημείο που δεν μπορεί κανείς να μετριάσει τον αντίκτυπο της ανεμογεννήτριας. Πρέπει απλά να φύγει από εκεί και να πάει κάπου αλλού. Θέλουμε να γίνει αξιολόγηση αντικτύπου και να δούμε τις επιπτώσεις τα μεταναστευτικά πτηνά και τις επιπτώσεις ε, σε ένα είδος χήνας το οποίο απειλείται με εξαφάνιση. Ούτως ή άλλως και έχει ενταχθεί στους σχετικούς καταλόγους. Θέλουμε παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς για το μέλλον ε, όλων των πτηνών που υφίστανται τον αρνητικό αντίκτυπο από τις ανεμογεννήτριες και να έχουμε σαφή εικόνα για τα, την αύξηση των ποσοστών θνησιμότητάς τους. Στρεφόμαστε λοιπόν προς τα εσάς και σας ζητούμε να μας βοηθήσετε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, να αξιολογήσουμε αρχίσουμε το μέγεθος, την ένταση, την οξύτητα του προβλήματος, να ε, έχουμε επιβολή της εκτίμησης ε, επιπτώσεων και να υπάρξει η καλύτερη υποπτία του βουλγαρικού κράτους της αντίστοιχης κυβέρνησης για να τηρηθούν και να γίνουν σεβαστές οι σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σας, ευχαριστώ Σας πολύ και η Επιτροπή, ο εκπρόσωπος Επιτροπής. Κυρία Ρέζεβα Κανάτης, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν έξι αναφορές που καλύπτουν ε, αρκετά θέματα. Θα συνοψίσω την κατάσταση αναφερόμενη στα προβλήματα. Ξεκινώ με την καλή άκρα. Από Από πλευράς εκπροσώπου αναφέροντος ή αναφέρουσας παρουσιάστηκε η κατάσταση ως έχει και η τοποθέτηση αυτή ε, λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με την Επιτροπή. Η διαδικασία επί έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, τον καθορισμό αυτή τη τοποθεσία στην καλή υπό την Οδηγία Προστασίας των Πτηνών και υπό τις οικονομικές δραστηριότητες ε, η δεύτερη πτυχή έχει ήδη συμμορφωθεί με το πρώτο τμήμα της ε, κατάστασης αυτή η Βουλγαρία. Για το δεύτερο τμήμα για τις οικονομικές δραστηριότητες η Βουλγαρία βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων σε σχέση με την απόφαση και την εξέταση μέτρων για την αποκατάσταση αυτής της ε, ε, κατάστασης πραγμάτων. Είναι σε επαφή με τις βουλγαρικές αρχές και παρακολουθεί του σύνεγγι στο θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να υπογραμμίσω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιβάλλει την λήψη μέτρων στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι μια ε, κατάσταση πραγμάτων που ισχύει και προτείνουν μέτρα τα κράτη-μέλη επί των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κρίνει αν είναι επαρκή ή όχι. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αναφέρεται στην αναφορά είναι η ε, δραστηριότητα όσον αφορά την, ε, την οικοδόμηση γύρω από ποταμούς και ε, λίμνες. Είχε ήδη κλείσει σε σχέση με το θέμα αυτό η εξέταση επειδή υπέβαλε μέτρα η, Ευρωπαϊκή, ε, η Βουλγαρία για την προστασία αυτών των τοποθεσιών. Και επιπλέον σύμφωνα με τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τακτά διαστήματα υποβάλλουν στοιχεία οι βουλγαρικές αρχές για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων. Τελευταίες πληροφορίες υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο φέτος και ανέφεραν ότι εξακολουθούν να ισχύουν αυτά όσον αφορά τα προβλεπόμενα οι ε, βουλγαρικές αρχές και έτσι εκ προημίου μας ενημέρωσαν σχετικά. Εξού και δεν βρήκε, δεν ε, εντόπισε κάποια παραβίαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευράς Βουλγαρίας όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα και έτσι και σε σχέση με αυτό το θέμα δεν ε, ε, δίνεται συνέχεια σε οποιαδήποτε άσκηση επί παραβάση. Αυτό σε σχέση με το, ε, την κατάσταση όσον αφορά τις, τα πλαίσια του 2007-2009 αναφέρονται μεταξύ άλλων σε σχέση με την ε, αναφορά 997-2007 και την ε, αντίστοιχη άλλη αναφορά του 2007 επίσης τη 1299. Το επόμενο πρόβλημα αφορά την μη επαρκή, τον μη επαρκή προσδιορισμό προστατευόμενων ε, περιοχών υπό την οδηγία για τους οικοτόπους σε σχέση με την ε, οδηγία 997 του 2007, την 1336 του 2008 και την 1519 του 2008 αναφορές. Όσον αφορά τον προσδιορισμό περιοχών και διατάξεων υπό την οδηγία για τα πτηνά και την προσπάθεια να καθοριστούν αυτές οι περιοχές από την Βουλγαρία με μια εξαίρεση όσον αφορά την περιοχή Ρίλα που έχει πολύ μεγάλη ε, σημασία για την προστασία αρκετών ειδών πτηνών μέσα σε έναν δασικό ε, οικότοπο. Λόγω της μη επάρκειας της Βουλγαρίας να συμμορφωθεί σε σχέση με αυτή την περιοχή αποφάσισε το Συλλογικό Σώμα των Επιτρόπων να ασκηθεί προσφυγή κατά της Βουλγαρίας για αυτή την περίπτωση. Όσον αφορά τον προσδιορισμό υπό την οδηγία οικοτόπων, Habitat, η κατάσταση είναι παρόμοια. Μπόρεσε να προσδιορίσει όλες ε, τις αναγκαίες ζώνες η Βουλγαρία με εξαίρεση κάποιες περιοχές ε, στα όρη Ρίλα. Και αυτό σε σχέση με την ε, εντεταλμένη έρευνα που βρίσκεται υπό εξέλιξη και βρίσκεται στην, ε, στις πρώτες φάσεις, ε, φάσεις της ε, Ολοκληρώντας, Ο μόνος προβληματικός χώρος ως πεδίο έγκυται στις, στα όρη Ρίλα για την Βουλγαρία. Οι υπόλοιπε ζώνες έχουν επαρκώς προσδιοριστεί είτε ως ζώνες ειδικής, ειδικής προστασίας είτε ως ζώνες κοινοτικής προστασίας. Επόμενο πρόβλημα είναι εδώ εκείνο το οποίο αφορά τις οικοδομικές δραστηριότητες στην παράκτια περιοχή της Μαύρης Θάλασσας στην ε, αναφορά 1299 του 2007 και την ε, αντίστοιχη 1336 του 2008 αναφορές. Ε, οι εξεταστικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων και σχεδίων έτυχαν αδειοδότησης από πλευράς Βουλγαρίας εκτός από μία περίπτωση που αφορά την εκαθάριση της κήτης ενός ποταμού. Γι' αυτό έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έπρεπε να τύχει συνέχεια αυτή η περίπτωση λόγω ελλειπών ε, ε, τεκμηρίων. Οι ε, επαφές με τις βουλγαρικές αρχές σε σχέση με αυτή τη διαδικασία, με αυτό το θέμα, κατέδειξαν ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν ένα μέτρο εκαθάρισης κήτης ποταμού για να αποφευθούν πλημμύρες. Έλαβαν όμως μέτρα για την προστασία της περιοχής οι αρχές ακόμα και την φύτευση και δημιουργία ειδικών προστατευόμενων περιοχών πράγμα το οποίο ε, ε, ε, έδωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έναυσμα να θεωρήσει ότι ήταν επακής η δράση από πλευράς Βουλγαρίας ώστε να κλείσει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον οι βουλγαρικές αρχές παρέσχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια έκθεση όσον αφορά την λήψη συνεχιζόμενων μέτρων και πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη αυτών των ζωνών όσον αφορά την Μαύρη Θάλασσα και όσον αφορά το τελευταίο τελευταίο προβληματικό θέμα όσον αφορά πολλαπλές αδειοδοτήσεις και δράσεις σε προστατευόμενες περιοχές την αναφορά 1336 του 2008 και την 1518 του 2008 και λόγω των ε, οικονομικών δραστηριοτήτων ε, που παραβίαζαν τις ε, κοινοτικές διαδικασίες στην περίοδο 2007-2009 στη Βουλγαρία. Οι, Ευρωπα... υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέδειξαν ότι πολλαπλά τέτοια προγράμματα είτε δεν υλοποιήθηκαν ή έληξε η άδειά τους σαν αποτέλεσμα εισαγωγής ε, από τις βουλγαρικές αρχές μιας πενταετούς ε, περίοδου μέσα στην οποία έπρεπε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αλλιώς θα έλεγε η αδειοδότηση. Βρίσκεται υπό εξέλιξη η διαδικασία και είναι πολύ πιο περίπλοκη και σύνθεση, σύνθετη σε σχέση με ε, άλλες αναφορές που αφορούν άλλες ζώνες ή περιορισμένου εύρους δραστηριότητες. Το επόμενο βήμα για την ανάληψη δραστηριοτήτων πρωτοβουλειών από πλευρά μα θα αποφασιστεί εν ευθέτω χρόνο σύντομα. Ευχαριστώ τώρα τον λόγο στου συναδέλφου. Κυρία Πιτέρα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά συμβαίνει το εξή. Στις ε, νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ένταξή τους δεν υπήρχε νομικό πλέγμα για το χαρακτηρισμό ή μάλλον για την τοποθέτηση αυτών των ανεμογεννητριών. Και δεν έλεγε τίποτα ο, η εθνική Δημοθεσία για το πού θα τεθούν αυτές οι ανεμογεννήτριες, αυτά τα ελληνικά πάρκα, ας πούμε. Αυτό έδωσε, οδήγησε σε πολλές διενέξεις. Το θέμα δεν έχει οικολογική διάσταση μόνο, αλλά και περιβαλλοντική και οικονομική, γιατί πολύ συχνά φτιάχναμε αυτά τα αιωλικά πάρκα κοντά σε μνημεία, ε, κοντά σε τουριστικές περιοχές ε, και αυτό στην πραγματικότητα οδηγούσε σε απώλειες για από τα οριστικά έσοδα, γιατί κανένα δεν θέλει να νοικιάσει ένα δωμάτιο όταν βλέπει αυτέ τι ανεμογεννήτριε. Επίση, δημιουργούσε πολλέ διαφορέ, πολλέ διενέξει ε, λόγω διαφθορά. Συχνά υπήρχαν πάρα πολλέ πιέσει από αυτέ τι επιχειρήσει που θέλουν να φτιάξουν τα, τα πάρκα αυτά ε, όπου να είναι και να πάρουν και άδεια. Πάντως υπήρξε δυνατότητα αλλαγή χάρη σε τη μεγάλη υποστήριξη που δόθηκε στο να κατασκευαστούν ε, αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να κατασκευαστούν οι ανεμογεννήτες παρόλα αυτά. Υπήρχε στήριξη του κοινού και επομένως οι επιχειρήσεις αισθανόταν ότι ήταν ε, στη σφαίρα του, της ατιμορρησίας και μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπήρξαν πάρα πολλές καταχρήσεις τελικά και εγώ θα ήθελα να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά όσο δεν έχουμε ξεκαθαρίσει όλες τις πτυχές της. Ε, σε, στο μέλλον θα προσπαθήσω να, να υποβληθεί ένα ερώτημα προς τη Βουλγαρία για να δούμε πότε θα εφαρμοστούν όλες οι, οι διατάξεις, ε, πότε όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει η Βουλγαρία θα τα κάνει και μόνο τότε μπορούμε να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Η Μάργαρετ. Εγώ ήμουν επικεφαλής μιας αποστολής ε, ε, διερευνητικής ε, στη Βουλγαρία πριν από λίγα χρόνια. Ετοιμάσαμε και μια έκθεση στο τέλος αυτής της αποστολής και είδαμε τα εξής πράγματα εκεί, στην αποστολή. Η στάση των αρχών ήταν ε, όχι και τόσο προστατευτική απέναντι σε αυτές τις λεγόμενες προστατευόμενες περιοχές. Παραδείγματο χάρη στα βουνά Ρίλα, αλλά και αλλού. Επομένως, δεν έχω και τόση διάθεση να πω ευθύ εξ αρχής ότι η Βουλγαρία, η Βουλγαρία συγγνώμη, έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατεύσει αυτές τις περιοχές, γιατί υπήρχαν άλλα συμφέροντα που είχαν προτεραιότητα σε όλη αυτή την ιστορία. Επίσης συζητήσαμε και το πού τοποθετούνταν αυτά αυτές οι αυτά τα αιωλικά πάρκα. Φυσικά θέλουμε αυτή την ενέργεια. Υπάρχουν τόσα θετικά στοιχεία. Και επιπλέον αυτές οι, οι ε, μπορεί κανείς να σταματήσει να τις λειτουργεί, να τις παροπλήσει πολύ εύκολα και να τις μετακινήσει σε άλλο χώρο. Δηλαδή, αν τη τοποθετήσει κανείς στην αρχή σε λάθος μέρο μπορεί να σταματήσει, μπορεί να τη μετα, μετα, μετακινήσει. Επίση, συχνά υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη και καλά να τις βάλει εκεί που έχει σκεφτεί στην αρχή. Μπορεί να υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Αν, α πούμε, εκεί που έχει σκεφτεί ότι πρέπει να μπουν ε, είναι χώρο ε, όπου φωλιάζουν τα πτηνά, ε, όπου υπάρχουν οικότοποι μεταναστευτικών πτηνών, μπορεί να τις βάλεις λίγο πιο πέρα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση για τον τόπο εγκαταστασής τους. Εάν, ας πούμε, εκτός από την αρχική πρόταση ότι θα, για την τοποθέτησή τους στο σημείο Χ, υπάρχει και εναλλακτική λύση. Μερικές φορές λόγω τεμπελιά, αμέλεια ή βλακεία δεν επιλέγει κανεί τη δεύτερη λύση που, που συχνά είναι καλύτερη από την, πρώτη, από την πρώτη λύση που σκεφτεί κανεί. Και στη Δανία είχαμε τέτοιους ιδιοκτήτε ε, ανεμογενετριών, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ υπερφύαλοι, επίμονοι, επέμεναν να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ μερικές φορές οι εναλλακτικέ περιοχές ήταν πολύ καλύτερες από, από το σημείο που είχαν σκεφτεί αρχικά ε, αυτοί. Ο κ. Μαρίνο. Details, uh, Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Να πω κάτι χρήσιμο. Ίσως και για μελλοντική συζήτηση, για οποιαδήποτε τέτοιου είδους αναφορά που αφορά τη Βουλγαρία. Όπως φαντάζεστε ε, κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού ολοκληρωτικού καθεστώτος οποιοδήποτε περιβαλλοντικό θέμα θεωρούνταν ότι είναι άμεση επίθεση εναντίον του, του κυρίαρχου συγγνώμη, ε, κομμουνιστικού κόμματος. Επομένως είχαμε πάρα πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα στη χώρα μου. Τα τελευταία 27-28 χρόνια άλλαξαν άρτητα τα πράγματα, αλλά υπάρχει σύγκριση ανάμεσα σε περιβαλλοντικέ ανησυχίε και όχι την πολιτική εξουσία, το πολιτικό ε, κατεστημένο, αλλά του επιχειρηματίε, τα οικονομικά συμφέροντα. Από τη μία το περιβαλλοντικό, από την άλλη το οικονομικό. Το οποίο είναι φυσικό βέβαια. Αλλά η έλλειψη παράδοση οδήγησε σε πολύ έντονε συγκρούσει. Έλλειψη παράδοση, δηλαδή προστασία του περιβάλλοντος και σχεδόν το 1 τρίτο της ε, επικράτειας της Βουλγαρίας είναι και στο μέλλον θα είναι ε, πολιτιστική κληρονομιά, φυσική πολιτιστική κληρονομιά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βούλγαροι πολίτες είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι η πολιτική εκπροσώπηση του Πράσινου Κόμματος ή των οικολόγων είναι πολύ αδύναμοι. Δεν υπάρχουν ούτε στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο και φυσικά δεν υπάρχουν ε, Βούλγαροι ε, ευρωβουλευτές οικολόγοι. Γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ενώ παραμένει ανοιχτή, ενώ αναφέρουμε Ρίλα Μπούφερ, Ηρακλή Κάντσια, τέτοια ονόματα, ας πούμε, βουλγαρικά ονόματα, όσο αντιχούν εδώ στο Κοινοβούλιο, θα υπάρχει πίεση στις βουλγαρικές αρχές στους ανθρώπους αυτούς που έχουν φυσικά τα συμφέροντά τους να προστατεύσουν και θα προσέχουν λιγάκι. Ε, δεν θα κάνουν τα χειρότερα, θα τους πιέσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι αναφορές και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και άλλες τέτοιου είδους αναφορές στο μέλλον. Yes, Margaret. Ναι. Μάργαρετ, ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα ότι στη Βουλγαρία είδα μια οργανωμένη κοινωνία των πολιτών που σφίζει από ζωή, με πάρα πολλή γνώση. Δεν ήταν άνθρωποι μόνο με απόψεις, αλλά και άνθρωποι που ε, στοιχειοθετούσαν επιστημονικά τις απόψεις τους, με σοβαρότητα. Όμως η γνώση δεν φτάνει στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση. Χρειάζεται μεγαλύτερη ορατότητα, καλά το λέτε. Να παραμείνει λοιπόν ανοιχτή αυτή η αναφορά και να απευθύνουμε την ερώτηση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έχουν κάνει. οι Βουλγαρία, η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών χρειάζονται τη στήριξή μας. Και θα πρέπει να πάμε το θέμα όσο πιο μακριά μπορούμε. Έχετε εξετάσει στην Επιτροπή τη στάση σας σε δεύτερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση Έχετε εξετάσει αν υπάρχει κάποια άλλη τοποθεσία διαθέσιμη. Εγώ προτείνω να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Η Πρόεδρος. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ακούμε τον κύριο Μαρινόβ να μας λέει ότι οι πράσινοι απουσιάζουν, αλλά εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να ε, προστατεύσετε το περιβάλλον. Αυτό είναι εξαιρετικό, εξαιρετική συνεργασία. Θα ήθελα τώρα να συνοψίσω, να προσπαθήσω να συνοψίσω λέγοντας τα εξή για τις διάφορες αναφορές. Ότι συμφωνώ πλήρως με τη Μάρκαρετ, με τον κύριο Μάλινοφ. Και λαμβάνοντας υπόψη αυτά που δεν είπε ή που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν κάποια επιχείρηματα υπέρ του να κλείσουμε την αναφορά και να προχωρήσουμε. 7, 13, 36 και 15-18 είναι αυτές που θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτές γιατί τα προβλήματα ε, παραμένουν και είναι έντονα. Θα, θα μπορούσαμε όμως να κλείσουμε τις αναφορές 1082, 640 και 12, 99 γιατί για αυτές έχει υπάρξει πρόοδος. Και σε γενικέ γραμμέ θα ήταν καλό να συντάξουμε μια ευρεία επιστολή γενικού περιεχομένου η οποία θα ε, συνοψίζει τι συζητήσει που είχαμε σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών, να απευθύνουμε την επιστολή τη σχετική στη βουλγαρική κυβέρνηση και να πούμε ότι ε, μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις και ότι παραμένουν τα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας. Μπορούμε αυτό να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Καλώς. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο. Έχετε δίκιο. Βιάζομαι τόσο που ε, ξέχασα να δώσω το λόγο στον αναφέροντα. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ να είστε πολύ σύντομος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Είναι σημαντικό οι αποφάσεις του δικαστηρίου να γίνονται σεβαστές. Ιδελαιώς καταραίει όλο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση παράβασης ε, της κοινοτικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ενέργεια, για το χρόνο που έχετε σπαταλήσει και που έχετε επενδύσει μάλλον σε αυτό το έργο. Είναι πολύ δύσκολα αυτά τα ζητήματα και δεν είναι εύκολο πάντοτε αυτό. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τη Μάργαρετ. Ας προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 21. Έχουμε τους αναφέροντες εδώ. Θα σας δώσω το λόγο για τρία λεπτά στο καθένα. Η Πιλάρ Μαρτίνεθ, ο Χωσέ Παύλο και ο Βιθέντε Τόρες και Άγχελα Παγκάλο. Τρία λεπτά ο καθένας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Με ακούτε? Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. αποφασίσαμε να συμπυκνώσουμε τις παρουσιάσεις των τριών σε μία παρουσίαση, αν μας το επιτρέπετε αυτό. Έχουμε φέρει μαζί μας έγγραφα που νομιμοποιούν και που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές της αναφοράς μας. Να πούμε καταρχάς ότι είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση για εμάς, όπως όλες οι υποθέσεις με τις οποίες ασχολείστε εσείς εδώ. Ωστόσο για εμάς είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε πρόσβαση στην Επιτροπή σας και ότι εσείς μπορείτε να μας ακούσετε. Όταν υποβάλαμε τα παράπονά μας, όταν ασκήσαμε τα αντίστοιχα ένδικα μέσα για τα θέματα που μας απασχολούν, για τους φυσικούς χώρους που εντάσσονται στο Natura 2000 ε, και στο δρυμό και στη ζώνη την προστατευμένη περιοχή στην ε, ε, ε, στην Αστούριας, Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε σε αυτό το αίτημα. Ξέρετε, μερικές φορές είναι οι πολίτες πολύ ευρωσκεπτικιστές γιατί πιστεύουν ότι είναι πολύ μακριά από αυτούς η Ευρώπη. Εμείς είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ακραδάντως ότι, ε, ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες απαιτούν εμεί να, δεν μπορεί να οι ευρωπαϊκές οδηγίες να απαιτούν να εμφανιζόμαστε συνεχώς ενώπιον δικαστηρίων για να δικαιωνόμαστε. Αυτά τα ένδικα μέσα ασκήθηκαν 97-99 και έγιναν δεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2004. Το άρθρο 4 της οδηγίας για τους βιότοπους ε, προβλέπει μία μέγιστη προθεσμία 6 ετών για να κηρυχθούν αυτές οι περιοχές ως ζώνη ειδική διατήρησης. Και στην Αστούρια αυτό έγινε με το διάταγμα του 2014 και το διάταγμα του 2015, διατάγματα που ακύρωσαν για δεύτερη φορά οι δικαστικές αρχές. Δηλαδή 20 χρόνια μετά από την ανακήρυξη των περιοχών σε ζώνες ειδική διατήρησης δεν έχουν ε, ε, κάλυψη νομική όλα αυτά και δεν έχουν γίνει δεκτά και ε, δεν έχουν εγκριθεί στο χάρτη όπου έχουμε τις διάφορες χρήσεις οικείς και στις σχετικές επιστολές που είχαν απευθυνθεί στην ε, κυβέρνηση είδαμε ότι είδαμε ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα. Ξέρετε, η Ισπανία είναι το 27% της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ κατά μέσο όρο τα άλλα κράτη συμβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια με 18%. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ανθρώπινοι πόροι με επαρκή γνώση για τα θέματα αυτά. 68.000 σελίδες είναι το υλικό τεκμερίωσης και είδαμε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι εργασίες επιτόπου. Δεν υπάρχει κατελάχιστον ορισμός γεωγραφικών αναφορών για να υπάρχει νομική ασφάλεια. Δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες, δεν υπάρχουν σχέδια προληπτικής δράσης, δεν υπάρχει ορισμός ειδικού προσωπικού. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν τηρείται η διαδικασία. Και δεν ισχύει το επιχείρημα της περιφερειακής διοίκησης δεν έχουν ε, εκπληρώσει η περιφερειακή διοίκηση ούτε καν τα μήνυμα προαπαιτούμενα ε, το, την προϋπόθεση των έξι μηνών. Και η περιφερειακή διοίκηση το αναγνωρίζει στο διάταγμα και λέει ότι θα έπρεπε να είχαν χωροθετηθεί αυτές οι περιοχές από πριν χρειάστηκε να προσφύγουμε στα δικαστήρια, στα οποία δικαιωθήκαμε και για δεύτερη φορά τα δικαστήρια κύρωσαν αυτό το διάταγμα. Όμως, ξέρουμε όλοι ότι όταν δεν τηρούνται οι κανόνες, αυτό σίγουρα επηρεάζει τα δικαιώματα των πολιτών. Πρέπει να φέρουμε αποδείξεις Ποια είναι καλύτερη απόδειξη από το γεγονός ότι ένα δικαστήριο μας δικαίωσε για δεύτερη φορά. Και σε 68.000 σελίδες δεν ε, υπάρχουν άλλες διαφορετικές επιστημονικές διαπιστώσεις. Θα ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, μελετήσει και να αναλύσει το ενδεχόμενο διορθωτικών δράσεων. και να αναθεωρήσει πλήρως τον κατάλογο, ο οποίος προτάθηκε πριν από 20 χρόνια και που 12 χρόνια μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να μην ισχύει στην Ισπανία. Δεν έχει ανακηρυχθεί η ζώνη ειδική διατήρησης και προστασίας σε αυτή η περιοχή και δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισής της. Και γιατί θέλουμε να αναθεωρηθεί. Γιατί αυτή η τοποθέτηση, ο λόγος που έκανε την Επιτροπή να εγκρίνει αυτά τα σχέδια τότε. Μπορεί να μην υπάρχει σήμερα. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν εκθέσεις που να τεκμηριώνουν αυτή την ανάγκη. Επομένως, το 90% ξέρετε της επικράτειας στην Αστούριας προστατεύεται και από το δίκτυο Natura και με άλλους τρόπους. Ουσιαστικά η εξαίρεση έγινε κανόνα στη δική μας αυτόνομη κοινότητα, στη δική μας περιφέρεια. Το 90% είναι προστατευόμενη περιοχή. Ουσιαστικά είναι διαστρέβλωση η γενικευμένη επέκταση, επέκταση χωρίς διακρίσεις μιας περιβαλλοντικής οδηγίας στο σύνολο της επικράτειας. Μια νομοθεσία και μια οδηγία η οποία εφαρμόζεται αλλού, παντού αλλού με πολύ επιλεκτικό τρόπο. Θα πρέπει να γίνει αυτή η αναθεώρηση ε, ε, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το πρώτο κόστος της διατήρησης είναι να αποζημιωθούν αυτοί που κομίζουν τη δική τους αδιοκτησία στο κοινό περιβαλλοντικό και εκτιμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού το 90% της επικράτειας εντάσσεται σε αυτά τα δίκτυα δεν υπάρχει κανένα είδου οικονομική αποζημίωση. Οικονομική αποζημίωση για του ε, ιδιοκτήτε, του μικροϊδιοκτήτες που είναι η ισχυρή πλειοψηφία των πληγέντων σε αυτέ τι επικράτειε, σε αυτά τα εδάφη. Και γι' αυτό το λόγο τα δικαστήρια κύρωσαν τα διατάγματα. Και υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, αυτό το οποίο ισχυριζόμαστε είναι ότι ε, καταστρατηγούνται θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, των κατοίκων που αναγνωρίζονται από τις συνθήκες και καταχειρώνονται. Υπάρχει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 27ης Τρίτης του 2009 σχετικά με την εξαιρετική αστικοποίηση της Ισπανίας και εκεί αναφέρεται ότι το δικαίωμα στη διονύδιο κτησία είναι θεμελιώδες και αναγνωρίζεται, κατοχυρώνεται στις συνθήκες της Ένωσης και η κατάπτωση και η καταστρατήγηση αυτού του δικαιώματος συνεπάγεται και η καταστρατήγηση και παραβίαση των ευρωπαϊκών συνθήκων. Υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία και δεν μπορεί κανείς να μπει σε αυτήν, ούτε καν ο ιδιοκτήτος της δεν μπορεί να μπει με εντολή της διοίκησης της δημόσιας και χωρίς καν να έχει πάρει αποζημίωση. Δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Είναι καταχρηστική δράση και την υφιστάμεθα από πλευράς της περιφερειακής κυβέρνησης της Αστούριας. Ε, πλήττονται τα δικαιώματά μας και ζητούνται εξηγήσει. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει αυτές τις διαδικασίες και να απαιτήσει να τηρηθούν και να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία ως Ευρωπαίοι πολίτες ερχόμαστε να επικαλεστούμε ενώπιον της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχουν διάφορα θέματα που αναφέρονται σε σχέση με την παρέμβαση του αναφέροντος. Πρώτον, ο προσδιορισμός όσον αφορά ζώνες και δίκτυο Natura 2000. Εδώ η οδηγία δεν καθορίζει ποια θα είναι, ποιο θα είναι το εύρος που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται από τα κράτη-μέλη στο δίκτυο Natura 2000. Δεν υπάρχει ούτε ελάχιστο ούτε ανώτατο κατόφλι γι' αυτό. Λέει η οδηγία ότι πρέπει να επιλέξουν αυτές ε, οι ζώνες τα κράτη-μέλη με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. Εξαρτάται λοιπόν αυτή η επιλογή από τον προσδιορισμό αυτών των οικοτόπων σε σχέση με την οδηγία και γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ισομερής ε, κατανομή. Και σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία σε σχέση με την Αστούρια, 27% σε σχέση με την επικράτειά της καλύπτεται από ζώνες ε, Natura 2000 ε, υπό την οδηγία για τους οικοτόπους και τους βιοτόπους και δεν έχουμε στοιχεία που να λένε και να αποδεικνύουν ότι αυτός ο προσδιορισμός έγινε με παραβίαση κριτηρίων. Δεύτερον, σε σχέση με την προστασία, προστασία αυτών των προσδιοριστικών ζωνών, έχουν την υποχρέωση τα κράτη-μέλη να θεσπίζουν και να υιοθετούν όλα τα αναγκαία μέτρα που είναι αναγκαία, ώστε να αποφευθεί η επιδείνωση των οικοτόπων και η όχληση ή επιδίνωση των βιοτόπων των ειδών και αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει περιορισμούς όσον αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες σε αυτές τις ζώνες. Η επιλογή λοιπόν αυτών των μέτρων επαφήνεται απόλυτα στη διακριτική ευχέρεια των αρχών των κρατών μελών. Μια άλλη πτυχή είναι η διαχείριση αυτών των ζωνών που ξεπερνά την πτυχή της απλής προστασίας. Η προστασία συνεπάγεται αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων. Όμως ε, η άλλη πτυχή συμπεριλαμβάνει και διατήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση αυτών των ζωνών. Εδώ λέει η οδηγία ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα διατήρησης ε, για αυτές τις ζώνες ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι διατήρησης που έχουν ε, τεθεί για κάθε ζώνη. Αυτά τα μέτρα μπορούν να έχουν πολύ διαφορετική φύση μεταξύ τους. Μπορεί να είναι προγράμματα διαχείρισης και σχέδια διαχείρισης, μπορεί να είναι μέτρα συμβατικά ή όσον αφορά το καθεστώς αυτών των περιοχών πάλι στη διακριτική ευκαιρία των κρατών μελών εφόσον αυτά τα μέτρα αντανακλούν τις οικολογικές ανάγκες αυτών των περιοχών και επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων διατήρησης όπως έχουν τεθεί στην Αστούρια συνειδητοποιήσαμε τα μέτρα διατήρησης πράγματι καθορίστη, είχαν καθοριστεί Ωστόσο πρόσφατα το Σεπτέμβριο 2016 υπήρξε κύρωση από πλευράς Ισπανικού Δικαστηρίου του διατάγματος όσον αφορά τον καθορισμό και τη θέσπιση μέτρων διατήρησης ε, για κάποιες ζώνες ε, του δικτύου Natura 2000. Αυτά είναι νέες πληροφορίες που έχουμε και θα τις λάβουμε υπόψη και θα τις συνεξετάσουμε συνολικά όταν θα έρθει η ώρα να αξιολογηθεί η απάντηση σε σχέση με τις διαδικασίες ε, επί παραβάση όσον αφορά την διαδικασία 2015 του 2003. Πρόκειται για μια διαδικασία επί παραβάση λόγω έλλειψης προσδιορισμού και ε, καθορισμού αυτών των ζωνών και ε, ε, ελλείψεις όσον αφορά τα μέτρα διατήρησης. Μια άλλη πτυχή είναι η χρηματοδότηση τα κονδύλια, χρηματοδότηση για την υποστήριξη όσον αφορά μέτρα διατήρησης ε, στις προστατευόμενες ζώνες. Εδώ ε, αντιλαμβανόμαστε ότι σε σχέση με τα όσα αναφέρονται, το Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για μέτρα της Natura 2000. Θα θέλαμε εδώ να υπενθυμίσουμε κάτι, ότι οι διατάξεις όσον αφορά την ανάπτυξη των μέτρων Natura συμπεριλαμβάνουν ρητά και προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την διατήρηση, προστασία και ε, διασφάλιση των οικοσυστημάτων που διασφαλίζουν ένα, την βιοπικιλότητα όσον αφορά τις προστατευόμενες ζώνες. Είναι το άρθρο 5 αυτό, αυτού του κανονισμού. Υπάρχουν και άλλα ε, άρθρα τα οποία αφορούν τις δράσεις και τις πληρωμές μέσα στο πλαίσιο της Natura 2000. Να χρησιμοποιείται αυτό το ταμείο για ε, την διατήρηση μέτρων και χρηματοδότηση μέτρων είναι ένα απόλυτα νόμιμο μέσο που επαφήνεται στην διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών όσον αφορά την συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις τους. Τελευταία τελική παρατήρηση όσον αφορά την προσπελασιμότητα σε αυτά τα στοιχεία. Η οδηγία 2003 κάθετος 4 θέτει την υποχρέωση στα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν την προσπελασιμότητα, την πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες για το κοινό και δεύτερον προοδευτικά να διαχέεται η πληροφόρηση όσον αφορά αυτά τα στοιχεία και ηλεκτρονικά. Τώρα, σαν συνέχεια της αξιολόγησης όλων των τεκμηρίων που κατατέθηκαν σε εμά στις υπηρεσίες μας, δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε οποιαδήποτε παραβίαση ή παράβαση παράβαση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές διατάξεις. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συμπεράνουμε, δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε κάποια παράβαση ή παραβίαση από τις Ισπανικές αρχές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα είναι η σειρά των Ευρωβουλευτών να παρέμβουν. Εσείς παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Σεσίλια. Η Αστούρης, όπως είδαμε, έχει 49 ζώνες προστατευμένες, 27% της επικράτειάς της ε, προστατεύεται, το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι εξαιρετικά αυτά στοιχεία. Φυσικά πρέπει να τα προστατεύσουμε αυτά τα, αυτές τις περιοχές και χρειάζεται μια ρύθμιση για τις ζώνες ειδικής σημασίας από περιβαλλοντική σκοπιά. Είναι ένα τρόπο για να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητά μας έτσι. Ακριβώς γι' αυτό ο νόμος και τα εργαλεία που τον εφαρμόζουν, όπως τα της ολοκληρωμένης διαχείρισης, πρέπει να εξασφαλίσουν την οικονομική αντιστάθμιση των πληττόμενων ιδιοκτητών, γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Και από την άλλη θα πρέπει να γίνει ένα σχέδιο διαχείρισης σε, για περιοχές που δεν μπορούν να συνεχίσουν οι κλασικές δραστηριότητες. Ε, και αυτό το σχέδιο δεν έχει σαν σκοπό για να λάβει κανείς ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αλλά θα πρέπει να γίνει περιβαλλοντική μελέτη για να δούμε κατά πόσο μπορούν να συνεχιστούν οι παραδοσιακέ δραστηριότητε. Στις απαντήσεις που μας έδωσε η Κομισιόν το 2015 και το 2016 δεν ε, προέκυψε ότι υπάρχει καμία παρατυπία σε αυτά τα εργαλεία ολοκληρωμένη διαχείριση. Φαντάζομαι και το ανώτατο δικαστήριο ε, όμως το νότο δικαστήριο του, της Αστούριας ακύρωσε το διάταγμα και δικαίωσε τους ε, προσφεύγοντες. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ο βασικός λόγος είναι, η βασική λόγη είναι δύο. Δεν υπάρχει καμία μνήμη για τη διαχείριση, ή μάλλον για αυτές τις δραστηριότητες. Σε πολλές περιπτώσεις Ε, υπάρχουν τεράστιες περιοχές, ας πούμε, ε, που είχαν αποκλειστική κτηνοτροφική δραστηριότητα, ας πούμε. Ε, υπήρχε μια μονοσήμαντη δραστηριότητα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Ε, και επιπλέον πρέπει να αναρωτηθούμε. Ε, όταν δεν λαμβάνουν ε, τις αποζημιώσεις οι διοκτήτες, για ποιο λόγο τις λαμβάνουν. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια έρευνα. Εδώ μιλάμε για δημόσιο χρήμα, το οποίο δεν φτάνει στα χέρια των δικαιούχων. Ε, φυσικά θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές αυτές, να, να στείλουμε μία επιστολή στην κυβέρνηση της Αστούριας για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και επιπλέον και μία στο Υπουργείο ε, Περιβάλλοντος. Και εν συνεχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, θα, θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία επί αντίον της Ισπανίας, αντίον της περιοχής, της αυτόνομης περιοχής, της Αστούριας πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ, η Ρώσα. Ευχαριστώ τους συντάκτες. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίε που μας έδωσε. Αυτό που είναι πιο σημαντικό στην αναφορά είναι ότι πολλές φορές Είπαμε στην Επιτροπή ότι δεν υπήρχε συμμόρφωση με ευρωπαϊκέ διατάξει, με ευρωπαϊκέ οδηγίε. Και πολλέ φορέ η Επιτροπή είπε όχι, ούτε το Δεκέμβριο του 2015, ούτε το Σεπτέμβριο του 2016, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση στη διαχείριση αυτών των χώρων του Natura 2000 στην Αστούρια. Ε, Επομένω, τα ε, Ισπανικά δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο τη Αστούρια Ε, καταργούν μία σειρά από διατάγματα. Επομένως κάτι δεν πάει καλά εδώ ε, και το λένε αυτό στην κυβέρνηση. Γιατί τα ισπανικά δικαστήρια, ε, εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα ισπανικά δικαστήρια και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι οι θεματοφύλακες, ας πούμε, της, του ευρωπαϊκού και ισπανικού δικαίου. Συμφωνώ με την Άχελα και με τους υπόλοιπους συμφωνώ, αλλά κυρίως με την Άγχελα, ότι χρειάζεται προστασία, αλλά όμως θα πρέπει να δοθεί επαρκής αποζημίωση στους δικαιούχους. Και δεν υπήρξε αποζημίωση ούτε μέσω των σχεδίων ε, διαχείριση. Νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Έδωσε νέα στοιχεία. Επιπλέον, περιμένουμε και τι αποφάσει του δικαστηρίου. Χρειαζόμαστε αυτό το χρονικό διάστημα, α πούμε, ε, ούτω ώστε και η Κομισιόν να εξετάσει το θέμα και να μα δώσει πληροφορίες για τα τεκτενόμενα. Ε, δεν έχω άλλους ομιλητές στον καταλογό μου. Πολύ σωστά είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όταν αξιολογηθεί το τι έχει γίνει από τις αρχές στην Στούρια και μια και δεν υπάρχει ε, παραβίαση ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα θέματα που αναφέρουν οι αναφέροντες στις αναφορές τους, αλλά, όπω όπως πολύ σωστά είπαν και οι δύο σα από την Ισπανία, απόκειται τώρα στην ε, Ισπανική κυβέρνηση να δώσει πλήρη αποζημίωση στους ανθρώπους αυτούς. Αυτό δεν είναι καθήκον ούτε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε τη Επιτροπή Αναφορών, αλλά καθήκον των Ισπανικών Αρχών. Να εξασφαλίσουν ότι η έλλειψη αποζημίωσης για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων που τους έχει επιβληθεί ε, δίδεται. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπέθρου προβλέπει πληρωμές αποζημίωσης, καταβολή αποζημίωσης και ενίσχυσης. Και στο άρθρο 30 προβλέπεται η δυνατότητα να δοθούν πληρωμές υπό το Natura 2000, ούτως ώστε να αντισταθμιστούν ε, για, τα περαιτέρω, για τα περαιτέρω έξοδα ας που έχουν, ή διαφυγόντα κέρδη που έχουν υποστεί οι κάτοχοι της γης, λόγω της πάυσης ή της αδυναμίας να ασκήσουν τις παραδοσιακές δραστηριότητε. Είναι μεγάλο πρόβλημα το γεγονό ότι δεν έχουν δοθεί αυτέ οι αποζημιώσει στου ανθρώπου που θα έπρεπε να τι είχαν ε, λάβει. Θέλουμε να αποζημιωθούν. Επομένω, να αφήσουμε ανοιχτέ τι αναφορέ μέχρι να λάβουμε απάντηση από τι Ισπανικέ Αρχέ για το θέμα αυτό. Πολύ ωραία. Αυτό θα κάνουμε και θα προχωρήσουμε. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο ξανά στου αναφέροντε, αλλά πολύ σύντομα παρακαλώ, εάν τον θέλετε. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστούμε. Καταρχάς, δεν υπάρχουν τεχνικές μελέτες ε, και τα 68.000 ε, σε 68 σελίδες αυτές του διατάγματος δεν υπάρχουν καθόλου αποδείξεις για αυτό το χαρακτηρισμό. Σε ό,τι αφορά τα κονδύλια του Γεωργικού Ταμείου, από αυτά τα κονδύλια δεν πήραμε δεκάρα. Το δικαστήριο λέει ότι εδώ καταγράφονται όλες οι οικονομικές δραστηριότητες από, από πολύ παλιά. Ας πούμε. Εδώ, αυτή είναι η μνήμη, ας πούμε. Ε, και όμως προβλέπονται κονδύλια από, την, από το Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπέθρου, τα οποία δεν τα λάβαμε ποτέ. Αυτά λένε αυτά τα έγγραφα. Αυτά τα έχουμε συνάψει στην αναφορά μας. Θα θέλαμε λοιπόν η αναφορά να παρέμβει για να εξετάσει πού πού πήγαν αυτά τα κονδύλια. Γιατί εμείς οι δικαιούχοι δεν ε, λάβαμε ούτε ένα ευρώ για ως αποζημίωση. Και σας διαβεβαιώ ότι έχουν παραβιαστεί διάφορα δικαιώματα, όπως, όπως ακόμα και η ελευθερία της κυκλοφορίας και, της, και Ε, δεν μπορείτε να μας ε, εμποδίσατε να κυκλοφορούμε, δεν μπορείτε να μας πάρει τις περιουσίες μας χωρίς αποζημίωση. Αυτό συμβαίνει στην Αστόρια όμως. Και εδώ ακριβώς ζητάμε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματά μας και για να απαιτήσει να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ επίσης και γι' αυτό. Είναι μια υποχρέωση αυτή σήμερα για τις αρχές στην χώρα σας και στην περιφερεια σας, σας να απελευθερώνονται κονδύλια σύμφωνα με τι νομικέ διατάξει και σύμφωνα με την οδηγία. Δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού. Αυτό όμω που μπορούμε να πράξουμε σε σχέση με τη δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι να αποστείλουμε μια επιστολή και να επισημάνουμε ότι ουσιαστικά παραμένουν αυτέ οι υποχρεώσει για αυτέ τι αρχέ και προσβλέπουμε σε γοργή απάντηση στις ε, ερωτήσεις μας. Και μέχρι να γίνει αυτό θα παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που ταξιδέψατε τόσο μακριά. Να ταξιδέψετε με ασφάλεια και να επιστρέψετε στην Ισπανία, στην όμορφη περιοχή σας και θα εξακολουθήσουμε να βρισκόμεθα σε επαφή. Τώρα έχουμε μια κοινή ανταλλαγή απόψεων για τη γνωμοδότηση για τα θέματα Μαρακές. Έχουμε μάγκα τη μία εισηγήτρια και τον συνάδελφο ως ε, συνεισηγητή. Έχουμε δέκα λεπτά, να είσαστε πολύ σύντομοι. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Το 2013 υπεγράφει η σύμβαση του Μαρακέσα. Όμως δεν μπόρεσε να αρχίσει να ισχύει σε σχέση με τα δικαιώματα τα πνευματικά ώστε στον οπτικοακουστικό τομέα να είναι δυνατόν να υπάρχει πρόσβαση στα βιβλία και στα προϊόντα αυτά. Σε σχέση με πολύ πρόσφατα δημοσίευσε μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα συγγραφικά δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα και όσον αφορά και τα, την οδηγία όσον αφορά την ε, ε, χρήση αυτών για άτομα που έχουν προβλήματα όρασης και είναι λαμβάνονται υπόψη ε, τα θέματα ε, και το πνεύμα της σύμβασης του Μαρακές όσον αφορά τη διασφάλιση ε, σε τέτοιου είδους προϊόντα για άτομα με προβλήματα όρασης. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν εδώ είναι το εξής. Να διατηρήσουμε την πρόταση αυτή όσον αφορά την πρόταση δηλαδή της Επιτροπής που θυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με όλα όσα προασπίζει η σύμβαση του Μαρακέσα και των συλλόγων και ενώσεων εξ ονόματος των ατόμων με προβλήματα όρασης και σε σχέση με τις αλλαγές όσον αφορά για παράδειγμα τις ρήτρες για την εμπορική εκμετάλλευση να μην υπάρξουν τέτοιες τροποποίησεις διότι αυτό θα ήταν αρνητικό σε σχέση με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που προτείνουμε είναι <clears throat> να μην ε, ε, έχουμε οποιαδήποτε τροποποίηση σε σχέση με το αιτιολογικό 11 διότι θα άλλαζε η κατεύθυνση των όσων θα προβλεπόντουσαν και σε σχέση με τις ε, δυνατότητες που υφίστανται όσον αφορά τα κράτη-μέλη να εντάσσονται μέσα στην, στα πλαίσια της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξού και η πρότασή μου είναι να διασφαλιστεί, να διατηρηθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις πολιτικές για τα άτομα με προβλήματα όρασης και για ε, μια ακρόαση που ε, ε, πρόκειται λοιπόν να γίνει σε σχέση με τις ενώσεις και συλλόγους εξ ονόματος αυτών των ατόμων. Σας ευχαριστούμε. Εσείς έχετε τον λόγο και θέλω να ευχαριστήσω και εγώ γι' αυτό και δεν θα μακρηγορήσω. Θα ήθελα να αναφέρω το εξής ο κανονισμός φυσικά είναι σημαντική υπόθεση διότι έχει ένα ευρύ πλαίσιο και πρέπει μέσα σε αυτό να μπορέσουμε να ενταχθούμε. Αν υπήρξαν κάποια προβλήματα, αυτό συνέβη επειδή τα κράτη-μέλη δίστασαν να υλοποιήσουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις που απορρέουν. Και εδώ έχουμε και θέματα ε, συμφερόντων και μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί όσον αφορά τα προτερήματα που θα συνεπάγεται η προσπάθεια αυτή για άτομα με προβλήματα όρασης. Η επικύρωση, η επικύρωση από τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να επιτευχθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και φυσικά κάτι μπορούμε να κάνουμε και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, εδώ η κατάσταση είναι η, η Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι σημαντικό και να βοηθήσει. Δηλαδή να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πρωτοβουλίες της και στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο κανονισμός αυτός να ολοκληρωθεί ταχύτατα. Και από πλευράς ε, Γιούρη ε, υπάρχει σύμφωνη γνώμη και συμφωνούμε, ίσως αυτό εκπλήξει κάποιους, το καλύτερο θα ήταν για τα άτομα με προβλήματα όρασης για την ανάγνωση στην Ευρώπη θα ήταν το δυνατόν νωρίτερα, πιο σύντομα να ολοκληρωθούν αυτά και να εγκριθούν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και με χαρά διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να εμπλακούμε και να ασκήσουμε την επιρροή μας ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και εξάλλου δεν έχουμε και πολύ χρονικό διάστημα, πολύ χρόνο που να απομένει στη διάθεσή μας και από πλευράς ε, εισήγησης, από πλευράς ε, ευθύνης για την ε, εισήγηση Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μου. Τρεις συγκεκριμένες προτάσεις υπό την ορολογία. Τι προτείνουμε εδώ σχετικά. Προτείνουμε η έννοια όσον αφορά διάθεση για άτομα με προβλήματα όρασης και τυφλούς το σύνολο της ομάδας αυτής των ατόμων να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία και η προστασία δεδομένων και αυτή να ενταχθεί σε αυτόν τον κανονισμό. Είναι το 216-279 Οδηγία 2002-58 όσον αφορά την προστασία δεδομένων. για όσους εμπλέκονται ε, ατομικά πρέπει αυτό να λαμβάνεται υπόψη. Και είναι σημαντικό να υπάρξει μια λύση αν υπάρξουν θέματα που δημιουργούν τριβές, ε, ε, κάποια προβλήματα, αν κάποιο όργανο για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι αρμόδιο για την επίλυση και διευθέτηση τέτοιου είδους διαφορών ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα διευθετούνται οι υποθέσεις αυτές και θα επιλύονται τα προβλήματα, ώστε να μπορέσει ο κανονισμός να λειτουργήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και να μπορέσει προς όφελος όλων των κρατών μελών να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί. Αυτά θα έπρεπε να είναι ο ανώτατος προτασικός μας στόχος και γενικά θα έπρεπε να γίνει η προσπάθεια τα, η σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου όσον αφορά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για άτομα με μειονεξίες, με ειδικέ ανάγκες να βρίσκεται πάνω πάνω στις προτεραιότητές μας. Σας ευχαριστώ. Εμείς είμαστε οι πρωτοπόροι και προπομπή όσον αφορά την πράσπιση της σύμβασης του Μαρακές. Δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές λοιπόν μεταξύ μας. Είμαστε συνενωμένοι στο στόχο και στην βούλησή μας αυτό να γίνει πραγματικότητα το νωρίτερο δυνατόν. Να σας πω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τροπολογίες προθεσμία για την κατάθεσή τους μέχρι 13 Δεκεμβρίου. Θα ψηφίσουμε στις 24 Ιανουαρίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στις 31 ε, Ιανουαρίου θα υποβληθεί η γνωμοδότησή μας ε, στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να δοθεί δυνατότητα τώρα στους συναδέλφους ευρωβουλευτές να παρέμβουν. Ωστόσο, μια και δεν έχουμε παρεκκλίνουσες θέσεις και απόψεις, ίσως να δώσουμε σύντομα τον λόγο απλά και μόνο στον εκπρόσωπο Μάρκο Γιορέλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Νομίζω ότι μπορώ πράγματι να τοποθετηθώ και στο πνεύμα της πρότασης και των στόχων που είναι κοινή όσον αφορά την αντιμετώπιση της νομοθετικής αυτής κατεύθυνσης δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω την προϊστορία και το, το, την ουσία της πρότασης. Γνωρίζω ότι τα μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής δραστηριοποιήθηκαν με ιδιαίτερο τρόπο ώστε να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη ώστε να αρχίσει να ισχύει η, συνθήκη, η σύμβαση του Μαρακές. Και γενικά με ικανοποίηση, ιδιαίτερη ικανοποίηση, παρατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωκοινοβούλιο γενικά καλωσόρισε χαιρέτησε τις ε, προτάσεις και την κατεύθυνση που επιθυμούσε η Επιτροπή, η Επιτροπή να ακολουθηθεί και θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική και πολύ εξειδικευμένη ταυτόχρονα αυτή η πρόταση και δεν ε, θα θέλαμε να εισαχθούν συγκεκριμένοι όροι, προϋποθέσεις, περιορισμοί ή άλλα στοιχεία εκτός από αυτά που είναι υποχρεωτικά από τη σύμβαση του Μαρακές για ένα τέτοιο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτων λεχθέντων λοιπόν καλωσορίζουμε, χαιρετίζουμε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωβουλή <clears throat> στόχευσε προς αυτή την κατεύθυνση και οπωσδήποτε γνωρίζουμε ότι εχθές υπήρξε ήδη μια πρώτη παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων Γιούρι και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε επίσης ε, το Συμβούλιο επιτελεί ε, ε, πρόοδο σε αυτό το χαρτοφυλάκιο και θεωρούμε ότι θα έπρεπε αν όλοι καθορίσουμε, παραμείνουμε πιστοί σε αυτές τις προτεραιότητες και στόχους, θα ενσωματωθούν όλα αυτά στη συζήτηση και στη στόχευση, ώστε να ολοκληρωθεί και να επικυρωθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο ήδη κατά την Μαλτέζικη Προεδρία, κατά το επόμενο εξάμεινο. Λοιπόν, είναι πρόθυμη να διευκολύνει όσο μπορεί αυτή τη διαδικασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί και ταχείς. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στις 12.30 και ξέρετε, είναι η τελευταία συνεδρίαση για φέτο τη κοινοβουλευτική μα επιτροπή. Η επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή Αναφορών θα διεξαρθεί στι 23 Ιανουαρίου 2017. Κάπως αμήχανα να αισθάνομαι να σας ευχηθώ καλά Χριστούμενα, Χριστούγεννα και θα σας ξαναδώ στους διαδρόμους. Υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου σας εύχομαι λοιπόν όλα τα καλά και εύχομαι ο επόμενος χρόνος να είναι και καλύτερος για όλους μας. Ευχαριστώ για σήμερα, θα είμαστε πάντα σε επαφή. Γεια σας.